Κυρίε Κυρίες και κύριοι, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή Ευστρική Αγορά ε, και Προστασία Καταναλωτών. Έχουμε αυτή την ε, δημοσιοκρόαση σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία για τα πυροβολά όπλα, για την οποία είχα τιμή, την τιμή να είμαι συγγητρία. να καλωσορίσω τους Ομιλητέ που έχουν έρθει από το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γαλλία, Ενωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και θα μας ε, φέρουν ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας. Έχουμε δημοσιεύσει πριν από μερικέ εβδομάδε και ένα άτυπο έγγραφο εργασία με το οποίο ζητούμε τη δική σα συμβολή σε πολλά τεχνικά ζητήματα και πραγματικά με έχει εκπλήξει ο όγκος πληροφοριών ε, και αντιδράσεων που έχουμε λάβει. Ένας από του σκοπού της σημερινή ακροαση είναι ακριβώς να καταγράψουμε ε, τα τεχνικά στοιχεία, τις τεχνικές πτυχές ε, της πρότασης, γιατί η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμπεριλάμβανε και μελέτη αντικτύπου. Γι' αυτό και δεν μπορούσε κανείς από την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει ε, ποιε θα ήταν οι πιθανές απροσδόκητες προεκτάσεις τη πρόταση, εφόσον δεν υπήρξε αξιολόγηση δικτύπου. Ελπίζω λοιπόν οι εμπειρογνώμονες να μπορέσουν να μας ενημερώσουν ε, για πιθανές ε, ε, συνέπειες της διατύπωσης της πρότασης της Κομισιόν, αλλά και για εμάς, ενδεχομένως να βοηθήσετε να βρούμε εναλλακτικέ προσεγγίσεις με νέες τροπολογίες. Η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Ξέρω ότι Κάποιοι σήμερα το πρωί δεν μπορούσαν να μπουν στο site. Εγώ μέσω Twitter έχω δημοσιεύσει το σύνδεσμο. Επομένω, ε, μπορείτε και εσείς να το αναπαραγάγετε για να ξέρουν όλοι πώς ε, να παρακολουθήσουν την συνεδρίασή μας ε, στο διαδίκτυο. Θα το βάλουμε και στο Facebook, αλλά θα μπορείτε να το βρείτε εκεί. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Φιλίπ Νόμπελς, μέλος της Επιτροπής Προβολών Όπλων που έχει σταθεί υπό την οδηγία. Για 25 χρόνια υπάρχει αυτή η οδηγία, που ξέρετε. Ο κ. Φιλίπ Νόβλης είναι το μέλος που εκπροσωπεί τη Γαλλία και έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι. Είμαι λοιπόν επικεφαλής ενός τμήματος για τα όπλα και τα κριτικά ε, στην, στο πλαίσιο της, ε, των αστυνομικών και δικαστικών αρχών μας. Και εδώ εξετάζουμε γιατί θεωρούμε σημαντικό να υπάρξει μια ε, αναδιατύπωση, μάλλον επανεξεργασία της οδηγίας. Γιατί ένα όπλο το οποίο είναι παράνομο στο παρελθόν μπορεί να ήταν στο νόμιμο πλαίσιο. Κάποια στιγμή δηλαδή από το νόμιμο κύκλωμα εξαφανίζεται. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν μια οδηγία που καλύπτει ε, αυτές τις νομικές διαστάσεις, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από το 1997 η Γαλλία έχει εντοπίσει ορισμένες ελλείψεις ε, για ζητήματα που είναι σημαντικά, όπως είναι ε, τα εξωτερωμένα όπλα και τα και τα άσφαιρα. Έχουμε λοιπόν ε, αυτή τον, τον παροπλισμό, του εξοδετερωσή τους ε, για ορισμένα όπλα και βλέπουμε ε, την διακίνηση τέτοιων όπλων που επέτρεψε στη συνέχεια την επαναχρησιμοποίηση αυτών των ε, όπλων με τις δραματικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. Στη συνέχεια, από το 8 μέχρι και το 2014, η ομάδα ΕΦΕ European Farm Experts, έχει εξετάσει ακριβώς αυτές τις νομικές ελλείψεις, τα νομικά κενά και έχουμε υποβάλει το 2009 στις αρμόδιες αρχές ε, ορισμένες ελλείψεις, ορισμένα παραθυράκια τα οποία θεωρούσαμε πολύ σημαντικά να διορθωθούν. Ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά την εξοδετέρωση αυτών των όπλων είχε υπάρξει αντίστοιχο αίτημα και ε, στις ε, αρχές αυτές που οδήγησαν το 2015 σε έναν κανονισμό. Όμως δεν έχουν επιληφθεί όλα τα ζητήματα. Οι επιθέσεις στο Παρίσι τον Ιανουάριο πέρυσι και τον Νοέμβριο ανέδειξαν ακριβώς αυτά τα κενά της νομοθεσίας και θέλουμε να υπάρξει λύση. Θα προσπαθήσω εν συντομία να θίξω ορισμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά τα εξωτερωμένα και άσφαιρα. Το γεγονός ότι δεν υπάγονται στην οδηγία τους επιτρέπει να ε, κυκλοφορούν χωρίς κανέναν περιορισμό. Δεν μπορούμε να πάρουμε πιο δεσμευτικά μέτρα γιατί δεν είναι πλέον όπλα, είναι απλώς αντικείμενα. Κατά τον ίδιο τρόπο, στην ε, οδηγία έχουμε συγκεκριμένα κανονιστικά κενά τα οποία θα ακολουθούν να υπάρχουν στην νομοθεσία, ιδίω σε ό,τι αφορά σημαντικές ε, έννοιες. Ποια είναι τα κύρια συστατικά ε, και τμήματα του όπλου. Ποια είναι τα κέρια αυτά τμήματα. Η ίδια αρχή ορισμένοι φορείς ε, ποια είναι τα, τα ουσιώδη συστατικά στοιχεία, ποια είναι τα άσφαιρα, ποια είναι ακριβώς αυτή η διαμεσολάβηση. Είναι μια μορφή εμπορίου που δεν ε, όμως ε, ε, προσδιορίζεται συγκεκριμένα. Όλα αυτά διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο και είναι σημαντικό να καλύψουμε αυτά τα στοιχεία. Αυτά επί των ορισμών. Ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό είναι η ανάγκη να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την ιχνηλασιμότητα των όπλων και όχι μόνο στις ε, ενδοευρωπαϊκές ε, κινήσεις. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία έλλειψη χνελεσιμότητας. Έχουμε έναν πρώτο ε, έλεγχο της χώρας στόχου που θα δεχτεί δηλαδή τα όπλα και υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο ε, κρατά ο εμπορευόμενος. Όμως η δημόσια αρχή δεν γνωρίζει πότε γίνεται αυτή η διακίνηση, ποιο όπλο μεταφέρεται και αν έχουν υπάρξει οι απαραίτητες άδειε. γιατί όλα αυτά τα έγγραφα τα κρατά στα χέρια του εμπορευόμενος. Ο ίδιος δηλαδή που κάνει αυτή τη μεταφορά. Και θεωρούμε σημαντικό η ανταλλαγή πληροφοριών για τις ενδοευρωπαϊκές κινήσεις να ρυθμιστεί και να βελτιωθεί η ρύθμιση της, γιατί υπάρχει μια σε εθνικό επίπεδο. Κάθε κράτος μέλος δηλαδή έχει έναν εθνικό, ένα εθνικό αρχείο για αυτά τα όπλα και τους αδιούχους όμως όταν ε, ένα όπλο φεύγει από μια χώρα και πάει σε άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξαφνικά σπάει εδώ η αλυσίδα της ειχνηλασιμότητας και αυτό είναι κάτι που διευκολύνει ε, το παράνομο εμπόριο. Η οδηγία λοιπόν έχει κενά όπως σας ανέφερα. Ένα από αυτά τα κενά είναι η επίσημη ε, ταυτοποίηση και καταγραφή του όπλου γιατί είναι απαραίτητο να έχουμε και τον κατασκευαστή, την αρχή, τον ε, χρονιά κατασκευή και ούτω καθεξής, αλλά στην εκκλονελασιμότητα του άπλου, όπλου, η επίσημη ταυτοποίησή του είναι και από την μάρκα, το μοντέλο, το, ε, τον αριθμό του ε, και το διαμέτρημά του. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στην οδηγία. Μετά, άλλο στοιχείο είναι και η διατήρηση των δεδομένων. Αυτή τη στιγμή είναι τα 20 χρόνια. Είναι όμως ε, εξαιρετικά σύντομο το χρονικό διάστημα και αν δείτε και με όλες αυτές ε, ε, τις επιθέσεις μπορούμε να έχουμε όπλα από το 1944, από, από πολύ παλιά μέχρι πιο πρόσφατα όπλα, επομένως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διατήρηση των δεδομένων και αυτά τα κενά είναι σημαντικά. Και αυτό φάνηκε και πρόσφατα από τις επιθέσεις του Ιανουαρίου πέρυσι στο Παρίσι. Είναι στοιχεία και κενά που γνωρίζουμε, όμως ε, έλαβαν δραματικές διαστάσεις γιατί τα όπλα τα οποία δεν είναι ούτε άσφαιρα με την έννοια της οδηγίας και του γενικού πρωτοκόλου ούτε εξωτερωμένα όπλα μπορούν να διακινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό επέτρεψε και την ε, δολοφονία στο εβραϊκό σούπερ μάρκετ. Τα όπλα αυτά έχουν κατακλείσει πολλές χώρες της Ευρώπης, πολύ σημαντικό πρόβλημα και θέμα. Ως, την αγορά, προς την αγορά πυρομαχικών, όπως και για ένα όπλο, το απλούστερο είναι δύσκολο να ταξινομήσουμε ε, ένα πυρομαχικό στην κατηγορία όπλων, διότι το ίδιο πυρομαχικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικά όπλα. Η ιδέα που είχαμε ήταν να πούμε ότι η αγορά του πυρομαχικού γίνεται μόνο από τη στιγμή που έχει νόμιμο τίτλο κατοχής του όπλου. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για άλλα αντίστοιχα πυροβόλα όπλα. Τα ακουστικά, τα όπλα κρότου είναι σημαντικά, τα τροποποιημένα επίσης ε, είναι σημαντικά, πρέπει να παραμείνουν στην αρχική τους κατηγορία. Ε, υπάρχουν όπλα που μπορεί να αλλάξουμε τον τρόπο ε, λειτουργίας τους, να αλλάξουν καθεστώς, να φύγουν στο εξωτερικό με εύκολο τρόπο μεταφοράς και μετά να ξανααλλάξουν και να επανέλθουν στο αρχικό τους καθεστώς ε, εκ των υστέρων. Για τις πωλήσει όπλων μέσω ίντερνετ Πρέπει αυτό να περιορίζεται μόνο στους επαγγελματίες που πρέπει να ελέγξουν για την δουλειά τους τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις πώληση. Αυτά και ευχαριστώ κυρία εισηγητρία. Ευχαριστούμε. Η συμφωνία είναι ως εξής παρεμβάσεις από τους τρεις επόμενους ομιλητές, 6 λεπτά ο καθένας και 20 λεπτά ερωταποκρίσεις και ερωτήσεις και απαντήσεις δηλαδή. Και μετά η δεύτερη ομάδα ομιλητών, πάλι 20 λεπτά ο καθένας, για 20 λεπτά συνολικά και μια άλλη σύνοδο ερωτήσεων απαντήσεων. Αν θέλετε λοιπόν να θέσετε ερώτηση παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι σας. Ο Πάνος θα τον κατάλογο. Πρώτος, Έντουαρτ Ήμπι, διευθυντής του Βασιλικού Μουσείου ε, Οπλισμού, Όπλων και Οπλισμού. I've been asked to speak. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τον ε, αντίκτυπο της οδηγία τα μουσεία και τι ιδιωτικέ συλλογέ. Για τα μουσεία στη Βρετανία θα μιλήσω, αλλά αυτό που θα πω ε, αφορά με διαφορετικό τρόπο και άλλα κράτη-μέλη φαντάζομαι. Η βασική ανησυχία μας, ε, και υπάρχουν και άλλες, είναι ο πιθανός ε, καταστροφικός αντίκτυπο στα ιδιωτικά πολιτιστικά προϊόντα που είναι όπλα και είναι μια κληρονομιά της ιστορίας και πηγή ενημέρωση για το μέλλον και έχουμε προτάσεις για το πώς μπορεί να, αποφευχθούν τα προβλήματα. Όπως έχει η κατάσταση, η 91 του 98 ε, μας ικανοποιεί. Τα προβλήματα αφορούν το άρθρο 2 και το άρθρο 6. Για το άρθρο 6 που αναφέρει από την αρχική οδηγία του 98 σε παχιά γράμματα ότι διαγράφεται το κομμάτι που είναι σε παχιά γράμματα και να αντικατασταθεί με αυτό, με αυτή την πρόταση. Η βασική λέξη είναι η λέξη απενεργοποίηση, δηλαδή απενεργοποίηση όλων των ε, όπλων κατηγορίας 1, στα, α στα μουσεία. Δηλαδή για να τα κρατήσουν ε, τα μουσεία πρέπει, που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αυτό δεν έχει σημασία για τα μουσεία. Εάν το αρχικό άρθρο 2.2 είχε διατηρηθεί. Γιατί στην παλιά μορφή του λέει τα εξή. Πάλι με το παχύ και σε πλάγι γράμματα στο τέλος. Η τροποποίηση ωστόσο διαγράφει την τελευταία πρόταση του 2.2 για τις με εξαιρέσεις μόνο για τις δημόσιες αρχές. Αν οι δημόσιες αρχές κρατήσουν, παραμείνουν στην εμβέλεια του αρχικού κειμένου, θα μπορεί να μην υπάρξει πρόβλημα, αν και θα πρέπει να δοθεί ορισμός τι σημαίνει στα αγγλικά τουλάχιστον, ο, τι εννοούμε με τον όρο public authority. Αλλά για να είναι συνεπή μεταξύ τους το 2 και το 6, η έννοια του, της δημόσιας αρχής, το, για τους οποίους δεν εφαρμόζεται η οδηγία, δεν μπορεί να είναι συνώνυμη με τα, τις δομές που ασχολούνται στο άρθρο 6 με τις συλλογέ των όπλων, αυτή, στις οποίες επιβάλλεται η υποχρέωση. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση για μας η οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα μουσεία να απενεργοποιήσουν τις, κατηγορι... τις συλλογές όπλων κατηγορίας Α. Τέσσερις είναι οι λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, πολιτιστική. Το όπλο είναι ένα ενεργό εργαλείο, δηλαδή έχει κινητά μέρη που περιέχουν το καινοτόμο, το ειδικό, το διακριτό σε σχέση με άλλα όπλα. Η απενεργοποίηση σημαίνει ε, ε ακροτηριασμός του στην πραγματικότητα. Αν, αν βγάλεις δηλαδή την, ε, ε, το, από το περίστροφο την, ε, ε θήκη, χάνει την ιδιαιτερότητά του. Θα οδηγήσει, στην, θα μοιάζει με μια καταστροφή τροποντινά. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Αυτό είναι το πρώτο επαναλαμβανόμενο πολυβόλο όπλο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι καθοριστική σημασία για την ιστορία του κόσμου. Άλλο παράδειγμα. Ένα ε, ημιαυτόματο όπλο. Μισό. a Του δώρο του Στάλιν στον Βρετανό πρέσβη του 1943. Επίσης έχει ιστορική και προσωπική σπουδαιότητα, πολύ μεγάλη. Μια δεύτερη πρακτική ομάδα λόγων, η απενεργοποίηση, κατα, καταστρέφει μια ενδυνάμει ζωτική σημασίας πηγή ενημέρωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να παράσχουν πληροφορίες και σε επιστήμονες και σε ε, αξιωματούχους της εθνικής ασφάλειας. Το Μουσείο Όπλων είναι εθνική πηγή στη Βρετανία έρευνας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Χρησιμοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις η τεχνογνωσία μας σε περιπτώσεις όπως από την ε, αντιμετώπιση του Άιρα, την, ε, το δικαστήριο των εγκλημάτων στην πρώην Ιγκοσλαβία κτλ. Αν χαθεί αυτή η δυνατότητα θα αυξηθεί η, ο κίνδυνος ε, ασφάλειας για τους πολίτες. Η τρίτη κατηγορία λόγων, η ανάγκη, η έλλειψη ανάγκης, ο κίνδυνος ε, για τη δημόσια ασφάλεια που, ε, που δημιουργούν τα προϊόντα αυτά στα μουσεία είναι μηδενικός. Τηρούμε μια σειρά πρότυπων που καλύπτουν τις ανάγκες ασφάλειας κάθε επίπεδου στην Βρετανία υπάρχει συμφωνία με την αστυνομία για τα επίπεδα ασφαλείας ε, των μουσείων που ελέγχουν την υλοποίησή τους. Επίσης υπάρχει ένα μητρό των συλλογών μας, ξέρουμε τι είναι, ποια είναι και που είναι. Στη Βρετανία ένα μουσείο για να έχει όπλα κατηγορίας Α πρέπει να πάρει ειδική άδεια από το κράτος και μια ειδική άδεια μουσείου που είναι δύσκολο να αποκτηθούν και περιλαμβάνουν μια σειρά σημαντικών κανόνων ασφάλειας. Εμείς είμαστε ένα πιστοποιημένο μουσείο με... όπου έχει κλαπεί ένα όπλο, αλλά δεν υπάρχει καμία, κανένα συσχετισμό μεταξύ της κλοπής όπλου και δημοκρατικών δραστηριοτήτων. Εμείς θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει έλεγχος. Η αφαίρεσή του, ωστόσο από τα μουσεία είναι διακριτικό. Αυτό, μιλά, αυτό αφορά ε, μουσεία που είναι ή δεν είναι ή υπό στατιωτικό έλεγχο. Αυτό δημιουργεί διακριτική αντιμετώπιση. Εγώ σας μίλησα για τα μουσεία και τους ορισμούς που χρειάζονται. Ένα μεγάλο κομμάτι της κληρονομιάς ωστόσο που μας απασχολεί, όχι στη Βρετανία αλλά αλλού, είναι στα χέρια ιδιωτών με την οδηγία όπως προκύπτει όλες ε, οι συλλογές, οι ιδιωτικές συλλογές θα καταστραφούν. Η πλειονομιά των προϊόντων, των όπλων είναι η ίδια, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε ανήκουν στο κράτος. Τι συστήνουμε τώρα, πολύ απλά. Πρώτον, την αποκατάσταση του άρθρου Δύο 2 ως είχε αρχικά που επιτρέπει σε ιδιώτες συλλέκτες και μουσεία να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις αυτές. Εναλλακτικά, μία τροπολογία στο άρθρο 2 που λέει τα εξή. πάλι παχιά και πλάγια. Οι εξαιρέσεις θα εφαρμόζονται σε συλλέκτες και οι συλλογές που ανήκουν στο δημόσιο και που ασχολούνται με, τη, με τα με τις πολιτιστικές και ιστορικές διαστάσεις των όπλων υπό την αίρεση της στήριξης από το κράτος, του, της νομοθεσίας του κράτους μέλους. Αυτή η τροποποίηση στην τροποποίηση θα μπορούσε να καλύψει όλους αυτούς ε, τις ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές που έχουν ιστορική σημασία ή πολιτιστική σημασία συλλογές όπλων. Θα τους επέτρεπε να έχουν όπλα που είναι λειτουργικά και ταξινομούνται στην κατηγορία Α. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο δεύτερος ομιλητής είναι ο δόκτωρ ε, Μάουρο Σιλβής, ο οποίος είναι διευθυντής της Ιταλικής Ένωσης Κατασκευαστών ε, Όπλων ε, ε, και Πυρομαχικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην ε, παρουσίασή μου θα ήθελα να εξηγήσω την άποψη της βιομηχανίας ε, σχετικά με την ε, τροπολογία της οδηγίας για τα όπλα λέγοντας ότι αυτή αφορά όπλα και επιθυμούμε να έχουμε την καλύτερη και νομοθεσία σχετικά με τα όπλα. Η ΑΝΠΑΜ ιδρύθηκε το 1980 στη Ρώμη και αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ε, όπλων, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για μια ΜΚΟ η οποία έχει και συμβουλευτικό ρόλο ε, στον ΟΗΕ αντικατοπτρίζει το 28% της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 50% ε, ε, όπλων πολυβόλων. Είναι μια ένωση η οποία ιδρύθηκε το 1976, η EEACS, Εκπροσωπούμε περίπου χίλιες εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στον τομέα και περίπου 150 κατασκευαστές ε, όπλων. Η επιρροή του τομέα μας λοιπόν ε, αφορά το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η παραγωγή ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια μονάδες ετησίως. Υπάρχουν 1.800 όπλα, ε, κατασκευαστές όπλων ε, και πυρομαχικών, 200 διανομής, 14.000 πολιτές και 300.000 συλλέκτες στην Ευρώπη. Οι αθλητικές δραστηριότητες εκπροσωπούνται ε, από 12 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι ε, τηρούν τους νόμους ε, ενώ η αγορά παράγει σε πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η δραστηριότητα αυτή λοιπόν υποστηρίζει 580.000 θέσεις εργασίας. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία λοιπόν χωρίζεται σε σε τρεις συνολικά οδηγίες, οδηγίες αυτήν του 91, 477 2008 κάθετος 51 η οποία ε, δέχτηκε τοπολογία και τέλος ε, τον κανονισμό 258-2012 ο οποίος εφαρμόζει το άρθρο 10 σχετικά με το πρωτόκολλο του ΟΗΕ για τα όπλα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι η Ευρωμαϊκή Ένωση εφαρμόζει πλήρως ε, το πρωτόκολλο του ΟΗΕ σχετικά με τα όπλα το ερώτημα τώρα είναι αν όλα τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία από το 2008 και έπειτα. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να μιλήσουμε για το χαρακτηρισμό μεμονωμένων σημείων του όπλου, το άρθρο 8 του πρωτόκολλου του ΟΗΕ, εφαρμόστηκε στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μέχρι το άρθρο 4 το και ορίζει ότι ο χαρακτηρισμός θα πρέπει να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του όπλου και η καταστροφή θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα το να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όπλο μετέπειτα. Τα μέλη κράτη λοιπόν, τα κράτη μέλη λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε όπλο κυκλοφορεί στην αγορά έχει ε, καταγραφεί με βάση αυτή την οδηγία ή ότι έχει ε, απενεργοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η, ε, η, η πρόταση της ε, Κομισιόν να τονίζει αυτή την ε, πρόταση ώστε να χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ένα μέρος του όπλου από την πλευρά του παραγωγού. Υπάρχει άλλη μια διαφάνεια η οποία εξηγεί τι ακριβώς είναι ο χαρακτηρισμός των μεμονωμένων μερών όμως έχουμε άλλον εκπρόσωπο εδώ, ο οποίος θα εξηγήσει καλύτερα το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ο χαρακτηρισμός των σημαντικών μερών είναι σημαντικό διότι ε, των ουσιαδών συστατικών ε, στοιχείων είναι σημαντικός διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε το χαρακτηρισμό στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν τα οποία δεν έχουν τέτοιο χαρακτηρισμό θα πρέπει να αναγνωριστεί με βάση τα άλλα κράτη-μέλη. Εδώ εξηγούμε ποια είναι τα ουσιώδη συστατικά στοιχεία. Έχουμε τα διάφορα μέρη που βλέπετε, μέρη που βλέπετε εδώ. Έχουμε εδώ ένα revolver, Ουσιώδη συστατικά ενός κυνηγητικού όπλου. Εδώ ένα ημιαυτόματο. Και ένα πυροβολό όπλο. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα όπλων ε, τα οποία έχουν διαφορετική διάμετρο, όπως ακριβώς υπάρχουν και χιλιάδες ε, μοντέλα αυτοκινήτων με διαφορετικές μηχανές. Ε, εδώ έχουμε μια φωτογραφία που μπορεί να σας κάνει να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι τα ουσιώδη συστατικά στοιχεία ενός όπλου ταιριάζουν και σε ένα άλλο. Χρειάζονται, χρειάζεται μεγάλη ειδίκευση για να μπορέσουμε να τα αποθηκεύσουμε σωστά και ε, ασφάλεια. Τώρα θα περάσουμε στα μη ουσιώδη συστατικά στοιχεία ε, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία ε, του όπλου και τα οποία μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν. Έχετε για παράδειγμα το σφυρί, την σκανδάλη, επιπρόσθετα υπάρχουν τα επιπλέον όπως είναι για παράδειγμα ε, ο, ε, το τηλεσκόπιο, ε, οι ο ορισμός των όπλων με βάση το πρωτόκολλο του ΟΗΕ ένα όπλο αφορά οποιοδήποτε όπλο το οποίο κρούει και το οποίο έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να κρούει μια σφαίρα ε, μέσω μιας έκρηξης χωρίς να συνυπολογίζουμε σε αυτό ε, ε, τις απομιμήσεις. Η απενεργοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία όχι, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά ένα όπλο. Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός του 2015, ο οποίος στηρείται σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι υποχρεωτικός από τον Απρίλιο του 2016 δεν θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθεί στην ε, ε, σκοπιά αυτής της ε, οδηγίας, στο πεδίο αυτή τη οδηγία. Τώρα όσον αφορά τα όπλα κρότου και συναγερμού, δεν ισχύει σε περίπτωση που μπορεί να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση και όλα αυτά δεν περιλαμβάνονται σε περίπτωση τα σηματοδοτούμενα, σηματοδοτούντα δεν συμπεριλαμβάνονται σε περίπτωση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και πάλι. Ε, τώρα ε, τα όπλα στην Αγερμού και τα σηματοδοτικά Ποιο είναι υπεύθυνο τώρα για αυτά, για την εφαρμογή της σωστής ε, νομοθεσίας. Β7, τα μη αυτόματα όπλα. Η υποκατηγορία Β7 συμπεριλαμβανόταν στο υπόμνημα 2 της οδηγίας του 1991. Τα τελευταία 25 χρόνια λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζήτημα τα οποία φορούν όπλα, τα οποία είναι αυτόματα και θεωρώ ότι σε όλη την Ευρώπη έχουμε βρει μια ισορροπία για αυτό. Επιπλέον όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, το καθένα τη δική του νομοθεσία για το συγκεκριμένο θέμα και αυτό νομίζω ότι είναι η πρώτη εναλλακτική που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και η κατηγορία Β7, Β7 ε, θα πρέπει να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε να βρούμε ε, ουσιώδη συστατικά μέρη του όπλου στην αγορά. Όμως μεταξύ των εναλλακτικών υπάρχουν πολλές άλλες εναλλακτικές οι οποίες θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να τις, να τις λάβουμε υπόψη μας ώστε να φτάσουμε μια συμφωνία και τη δημόσια ασφάλεια. Η μετατροπή τώρα των αυτόματων όπλων όσον αφορά την ε, μετατροπή αυτόματων όπλων θα ήταν αναγκαίο να επιβεβαιώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκές κατευθυντήριες για την σωστή από στρατικοποίηση των όπλων. Ε, θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν αυτά τα όπλα θα πρέπει να απαγορευτούν ή αν υπάρχει ένας επιστημονικός τρόπος να τα διαχειριστούμε και να έχουμε μια ασφαλή κατευθυντήριο για αυτό. Κλείνοντας, ε, τα όπλα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται με βάση ένα ουσιώδες θετικό στοιχείο τους, ώστε να αποφεύγουμε τα παραθυράκια και τα λάθη, σχετικά ε, με τα όπλα θα πρέπει ε, να τα απενεργοποιημένα να μην μπορούν να επανέλθουν και ε, να μην συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της οδηγίας τα συναγερμού και σηματοδοτικά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο της οδηγίας δεδομένου ότι τηρούν το άρθρο 1 της οδηγίας 2008-51 και οποιαδήποτε συστατικά τα οποία δεν περιλαμβάνουν ένα μία, περιλαμβάνουν ένα μία απενεργοποιημένο ε, συστατικό στοιχείο ε, θα πρέπει να ε, μπουν στην κατηγορία. Είναι σημαντικό να έχουμε ευρωπαϊκές οδηγίες, μια ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την αποστρατικοποίηση ως μια εναλλακτική από του να τα απαγορεύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να θυμίσω τους... Ε, ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι άμα έχετε κάποιες ερωτήσεις, απλά σηκώστε το χέρι σας για να καταρτήσουμε τη λίστα. Κρατήστε το χέρι σας όρθιο όσο σημειώνουμε τα ονόματά σας. Ακολουθεί στη συνέχεια ο υποδιευθυντής της ομάδας έρευνας ε, και πληροφορία σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, η συζήτηση για την πρόταση οδηγίας ε, Κάποιε φορές περιορίζονται συγκεκριμένα στοιχεία μόνο. Μάλιστα η πρόταση αυτή έφτασε ακριβώ πριν, μετά τι επιθέσει στο Παρίσι ε, και παρουσιάστηκε ω μια πρόταση κατά καταπολέμησης τρομοκρατία, το οποίο δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα. Όπω ανέφερε η Φίλη Νόβουλο προηγουμένω. Ε, δεν έρχεται από το πουθενά αυτή η πρόταση οδηγία. ήταν αποτέλεσμα μια μακροχρόνια διαδικασία. Και είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο να ρυθμίσει την αγορά νόμιμη αγοραπολισία. Και να θέσει στεγανά μεταξύ του της νόμιμης και παράνομης αγοράς. Προσπαθεί να εφαρμόσει μέσα διατάξεις του Διεθνούς Πρωτοκόλλου του ΟΗΕ για τα πυροβολα όπλα, καθώ και την κάλυψη ορισμένων νομικών κενών που υπάρχουν και έχουν προκύψει από αξιολογίες που έχουν γίνει κατόπιν αιτήματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής τελευταία χρόνια. Ω προς αυτό, η πρόταση οδηγίας συμπεριλαμβάνει σημαντικό αριθμό διατάξεων που είναι χρήσιμε και απαράδεκτε σε ό,τι αφορά ας πούμε, το χαρακτηρισμό, την ειχνελεσιμότητα των διαδικτυακών πωλήσεων, αλλά και πολλά στοιχεία όπου γύρεται ζήτημα σε φορά το εύλογο και το εφικτό των προτάσεων και μάλιστα κάποιες φορές φαίνεται ότι θα μας οδηγήσει αυτές τα αποτελέσματα η πρόταση. Ένας καλ... Οι νέοι ορισμοί ε, της μεσητείας και της μεσολάβησης είναι πιο σαφείς η συμπερίληψη σιγαστήρων και αντίστοιχων συστατικών είναι κάτι το θετικό. Όμως αυτοί οι σιγαστήρες δεν θα πρέπει ε, να μπουν κατευθείαν στην κατηγορία των ε, ουσιοδών μερών. Είναι ε, συμπληρωματικά μέρη. Και πρέπει όλα αυτά να εξεταστούν στο πλαίσιο της, του χαρακτηρισμού, του marking και εν γέννη μια, ένας εύρωστος ορισμός ε, και των συμπληρωματικών μερών είναι απαραίτητη γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος που παίζουν και αυτά τα μέρη και στο παράνομο εμπόριο όπλων. Σε ό,τι φορά το άρθρο 2.2 είναι κάτι το οποίο συζητείται ευρέω. Κατά τη γνώμη μας η συμπερίληψη των συλλογών, συλλεκτών και των ιδιωτικών ε, μουσείων είναι κάτι το προφανές. Ε, δεν πρέπει εδώ να αμφισβητήσουμε την καλή πίστη και την ακαιρεότητα των ε, συλλεκτών και των μουσείων. Περισσότερο είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας. Και οι χώροι που έχουν πολλά όπλα θα πρέπει να επάγονται σε αυστηρούς και επαρκείς κανόνες για να μην επιτρέπεται η μεταφορά αυτών των όπλων προς το παράνομο περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία Α, για πολιτισμικούς και ιστορικούς λόγους, ε, είναι λογικό και αποδεκτό να έχουν πρόσβαση τα μουσεία και οι συλλογές, αρκεί να έχουν και επαρκή μέσα ασφάλειας. για να αποφύγουμε τη σκόπιμη ή και μη σκόπιμη διαρροή αυτών των όπλων προς το παράνομο κυκλώματα. Εάν υπάρχουν ιστορικοί και πολιτισμικοί λόγοι, πρέπει πάντα να ε, προσδιορίζονται πολύ ξεκάθαρα και να περιορίζονται. Πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθο. Σε ό,τι αφορά τα εξουδετερωμένα όπλα, η πρόταση οδηγία συμπεριλαμβάνει ε, Συγκεκριμένε ασυνέπειε κατά τη γνώμη μα. Αν η συμπερίληψη αυτών των όπλων είναι κάτι το θετικό, μπορούμε από την άλλη να, να ρωτηθούμε κατά πόσο τα όπλα τη κατηγορία Α όταν εξωτερωθούν παραμένουν σε αυτήν την κατηγορία Α. Και έτσι υπάρχει μια ασυνέπεια, ενώ έχουμε υιοθετήσει κανονισμό για τα κοινά μέτρα εξουδετέρου απενεργοποίηση. Μπορούμε να πούμε ότι οι νέοι κανόνες είναι ανεπαρκείς τότε θα πρέπει να εξετάσουμε και τον κανονισμό. Εναλλακτικά θα πρέπει στην κατηγορία Α να βάλουμε μόνο τα ε, όπλα ε, κατηγορίας Α που έχουν εξωτερωθεί και δεν καλύπτονται από τον κανονισμό ή έχουν εξωτερωθεί πριν από την ημερομηνία θέση σε ισχύ του κανονισμού. Και έτσι ε, ακολουθούν λιγότερα, λιγότερα αυστηρούς κανόνες. Και όπως και να έχει, για σκοπούς συχνελεσιμότητας των απενεργοποιημένων, το σύνολό τους θα πρέπει ε, τουλάχιστον αναφέρονται ως ε, όπλα κατηγορίας Γ. Ένα άλλο ζήτημα ακανθόδες σε ό,τι αφορά τα μη αυτόματα ε, που χρησιμοποιούνται όμω για μη στρατιωτική δράση. Όταν αυτά βρίσκονται στα όπλα που υπάρχονται σε άδεια, η αδειοδότηση προκύπτει από την μορφή του όπλου. Όταν περνούμε στην ε, κατηγορία των απαγορευμένων όπλων, τότε ε, βλέπουμε τους περιορισμούς ε, αυτής της προσέγγισης που πλέον δεν είναι εφαρμόσιμοι. Έχουμε πολλά όπλα τα οποία αδειοδοτούνται βάσει μόνο της όψης τους. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος αριθμός των όπλων α7 να μην δηλώνονται και να περνούν έτσι στο παράνομο κύκλωμα και πέραν των του εύρους δράσης των ε, δημοσίων αρχών. Αυτό συνέβη και στο Βέλγιο. Πρέπει να δούμε για ποιους λόγους αυτή, έχει γίνει αυτή η αλλαγή κατηγορίας. Ε, σε ποια ουσιαστικά στοιχεία βασίζεται αυτή η απόφαση και ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ασφάλεια των κατοίκων. τώρα αν θέλουμε να θυμώσουμε, να, να χάσουν ψυχραιμία τους οι οι ερασιτέχνε, τότε το, το έχουμε καταφέρει. Όμως πρέπει να δούμε και τις προεκτάσεις σε ό,τι αφορά τη μετατροπή των ημιαυτομάτων σε αυτόματα. Πρέπει να βασιστούμε σε σε κανόνες σε ό,τι αφορά τον ε, περιορισμό ε, συγκεκριμένων ε, τεχνικών προδιαγραφών. Πρέπει να πούμε επίσης ότι τα ημιαυτόματα της κατηγορίας Β7 ε, πλέον δεν είναι μετατρέψιμα. Είναι πολύ δύσκολο να μετατραπούν από τους κατασκευαστές, όπως έχει γίνει για πολλά μοντέλα που βρίσκονται στην κυκλοφορία. Αυτό μπορεί να το πιστοποιεί και ένας ανεξάρτητος φορέας, όπως ισχύει ε, και με τον αντίστοιχο φορέα στις ΗΠΑ που ελέγχει και τα όπλα. Τώρα, οι εξαποστάσεις πωλήσει. σε ό,τι αφορά τις ε, ισχύουσες ε, τάσεις, σε ό,τι αφορά την ε, πώληση όπλων μέσω διαδικτύου, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν και κάποιες φορές γίνονται εκτός νόμιμου πλαισίου. Το να απαγορεύσουμε τις πωλήσει διαδικτύου πέραν των μεσητών και αντιμεσολαβητών είναι κάτι το θετικό. Θα πρέπει να αναρμονίσουμε τις πρακτικές. Όμως όλα αυτά δεν φτάνουν αυτό το μέτρο μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο μόνο αν συνοδεύεται και από αυστηρό έλεγχο των εξαποστάσεων αγορών, έλεγχο των αγοραστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ακολουθούν ε, τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό θα αποτελούσε πολύ σημαντικό κενό αν είχαμε πόπλα τα οποία απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν πιο εύκολα να επαναργοποιηθούν, ξαναβρεθούν με κάποιον τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια λύση θα μπορούσε να είναι τα όπλα τα οποία έχουν αγοραστεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάντα να ακολουθούνται από επαλήθευση της ταυτότητας του αγοραστή και να υπάρχουν και απαραίτητες άδειε μέσω της αρμόδιας δημόσιας αρχής. Και εδώ μιλώ ε, για έναν έλεγχο που αποτελεί αυτό σκοπό. Πρέπει όμως να έχουμε συγκεκριμένους ε, ε κανόνες στην οδηγία που να έχει τα λιγότερα δυνατά νομικά κενά και να μην επιτρέπει και να μην διευκολύνει ε, την παράνομη διακίνηση. Τα προβλήματα της ε, μετατροπής ε, και τη επανενεργοποίησης των όπλων δεν τα φανταζόμαστε από μερικά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα αναλαμβάνει δράση για να καλύψει αυτά τα κενά. Σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο υπάρχει αυτή η τάση. Και είναι απαραίτητο να ενεργήσουμε προδραστικά και ολοκληρωμένα, ούτω ώστε οι κακόπιστοι να μην εκμεταλλευτούν ε, τις ε, συνέπειες της οδηγίας. Να κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Uh, Υπάρχει χρόνος για 20 λεπτά ερωτήσεων. on the list, but because I'm the Είμαι και εισηγήτρια και θα θέσω και εγώ μια ερώτηση. Υπάρχει κανείς άλλος πέραν αυτών που ανέφερα που θέλουν το λόγο. Που θέλουν να θέσουν ερώτηση δηλαδή. Για τον πρώτο ομιλητή. Τι ακριβώς ζητήσετε για το θέμα της ιχνηλασιμότητας και των μητρώων. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλες οι χώρες έχουν υποχρεώσει σήμανσης. Προτείνεται, λέτε μάλλον ότι το σύστημα των ε, ε, μητρών δεν λειτουργεί ή δεν εφαρμόζεται σωστά. Το δεύτερο ερώτημα για τα μουσεία. Για τα μουσεία το καταλάβει. Για τους συλλέκτες γιατί καίγονται τα μουσεία. Κύριε Σίλβης, Εσείς λέτε ότι η σήμανση πρέπει να αφορά ένα ουσιώδες στοιχείο κάθε ε, όπλου, αλλά η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει σήμανση κάθε ουσιώδος συστατικού στοιχείου. Αυτό είναι η πρώτη μου ερώτηση εμένα, αλλά θα αφήσω τους αδέρφους να θέσουν τις ερωτήσεις τους, η Άννα Μαρία. Είμαι σκιώδη συγγήτρια για το ΕΛΚ και καλωσορίζω ιδιαίτερα την ακρόαση αυτή διότι μπαίνουμε στην ουσία της δουλειάς που χρειαζόμαστε, ε, την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία ειδικών. Και τον κύριο Ήμπεϊ, συλλέκτες και μουσεία. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Πότεβα, το θέμα της ασφάλειας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου όπλα συλλεκτών χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς ή έγιναν μπήκαν στην παρανομία. Η ασφάλεια στα μουσεία και τις δημόσιες συλλογές είναι κατά την άποψή σας επαρκής. Ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι η απαγόρευση των όπλων κατηγορίας Α από μουσεία και ιδιώτες ε, είναι κάπως ε, παρατραβηγμένη, πολύ παρατραβηγμένη. θέλω να καταλάβω περισσότερο. Μετά, οι ιδιωτικές συλλογές. Γιατί αριθμό όπλων μιλάμε. Για τον κύριο Σίλβης, ε, περισσότερο για το θέμα εφαρμογή. εφαρμογής, η παρέμβασή σας ε, έλεγε δεν χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες, αλλά καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της σύμβασης του ΟΗΕ. Ποια, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εφαρμογής, πού θα έπρεπε να στρέψουμε τη δουλειά μας. Τον κύριο Ποτεβάν. Εξ αποστάσεως πωλήσει. Δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά τέλος πάντων σέβομαι την εμπειρία σας και θέλω να ξέρω περισσότερο. Γιατί πρέπει να απαγορευτούν οι εξ αποστάσεως πωλήσει. Υπάρχει ήδη η μαύρη αγορά. Μέσω του σκοτεινού διαδικτύου. Η, ε, ο αγοραστής και ο πολιτής που έχουν άδεια πώληση και αγοράς αντίστοιχα αυτό κάνουν. Γιατί να απαγορεύσει την εξαποστάσεω πώληση γενικά. Αυτό θα πλήξει τα άτομα που ζουν στην Ήπεθρο. Η οδηγία αφορά τα νομίμως ε, τα όπλα που υπάρχουν με νόμιμο μέσα στην κατοχή κάποιου. Γιατί να μην αγοράσει κάποιο εξ αποστάσεω νόμιμα ένα όπλο που χρησιμοποιεί, θα το χρησιμοποιεί στον ελεύθερο χρόνο του. Δηλαδή η επιχειρηματολογία σας δεν μου έγινε κατανοητή. Θα ήθελα να ακούσω κάτι περισσότερο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση της Επιτροπής απαγορεύει πλήρως τα όπλα, την ιδιωτική κατοχή όπλων κατηγορία Α. Στην υφάρχουσα οδηγία υπάρχουν, ε, υπάρχει απαγόρευση με κάποιες εξαιρεσει για μουσεία και συλλέκτες. Μιλούμε για όπλα που έχουν μεγάλη ιστορική αξία. Η αναδρομική απαγόρευση κατά συνέπεια πρέπει να είναι θεμελιωμένη. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι η απαγόρευση και μη αναδρομική να είναι θα σκοτώσει την σχετική αγορά και θα μειώσει σημαντικά την αξία των όπλων. Η Επιτροπή έχει πει πολλές φορές ότι οι συλλέκτες όπλων είναι πηγή παράνομων, παράνομης Αυτό είναι προσβλητική δήλωση εκτός αν τεκμηριωθεί. Στη χώρα μου, τη Φινλανδία, υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός νόμιμων αυτόματων όπλων σε ιδιωτικές συλλογές. Συνήθως είναι οπλοπολιβόλα ή, ή, ή μη αυτόματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Βάσει των εθνικών αρχών τα όπλα αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ για εγκληματικές δράσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι με εμπειρική γνώση είναι πρόβλημα στην Ευρώπη τα ιδιωτικής κατοχής αυτόματα όπλα ή μήπως προσπαθεί η αυτοματα του δευτερου παγκοσμιου πολεμου βασει των εθνικων αρχων τα οπλα αυτα δεν εχουν χρησιμοποιηθει ποτε για μήπω προσπαθεί η ερωτηση μου λοιπον ειναι με εμπειρικη γνωση ειναι προβλημα στην ευρωπη τα ιδιωτικη κατοχη αυτοματα οπλα η μηπως προσπαθει η κομισιον να διορθώσει κάτι που δεν έχει χαλάσει. Κύριε Γιάχασάρη. Ευχαριστώ. Κάποιος από τους ειδικού σας δήλωσε ότι η συζήτηση για την οδηγία ήταν κάπως μινιμαλιστική. Δεν θυμάμαι άλλη οδηγία όπου είχαμε κάνει τόσες πολλές συζητήσεις. Και ευχαριστώ τη Βίκη Φόλ γιατί έδειξε μεγάλη υπομονή. Έκανε αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα. Ο στόχος είναι να αποφύγουμε την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος και το λαθρεμπόριο όπλων. Σημαντικός στόχος. Αυτό που θέλω να ακούσω από τους ειδικού είναι αν υπάρχει μια κάποια ευαισθησία για την διαφορετική κατάσταση από κράτος σε κράτος και την ανάγκη διαφορετικών λύσεων ένα παράδειγμα, το είπε ο προηγούμενο ομιλητή, ε, προφανώς ο στόχο τη οδηγία δεν, δεν είναι να αντιμετωπίσει την άμυνα μια χώρα. Στην περίπτωση της Φιλανδίας, για παράδειγμα, δεν καταλάβουμε ότι η άμυνα της Φιλανδίας στηρίζεται σε μια ευρείας βάσεως ε, χρήση εφέδρων της χώρας που έχουν όπλα ε, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Η πρόταση της Επιτροπής για το παράτημα 1 που δίνει τις κατηγορίες των όπλων και την κατηγορία των απαγορευμένων όπλων μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου θα τίθεται σε κίνδυνο η άμυνα μιας χώρας. Ελπίζω να το καταλάβουν. Μπορεί να είναι μικρή η λεπτομέρεια, αλλά καταλάβετε ελπίζω ότι αν ξέρετε την ε, ύπεθρο, την επαρχία σε πολλές χώρες, νέοι και νέες πια έχουν ως χόμπι το κυνήγι και ε, ανήλικοι πηγαίνουν στο δάσος να κυνηγήσουν. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τη δυνατότητα αυτή, να μην βάλουμε ένα όριο 18 που θα εμποδίσει τους 16χρονους ή τους 17χρονους από το να βγουν στο κυνήγι. Tästä Συνολικά ελπίζω και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα από την ε, συζήτηση των θεμάτων που τέθηκαν εδώ. Ευχαριστώ. Merci Madame la Présidente. Je voulais remercier les différents intervenants. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους ομιλητές. Πολύ σωστά τα όσα είπαν, αλλά πρέπει να επιθυμίσουμε τα εξή. Ε, Ιδίω η ψευδή αντίληψη με βάση την οποία έχουμε μια αυστηρή διάκριση μεταξύ ε, της νόμιμης ε, και πολύ καλής αγοράς και της παράνομης αγοράς που είναι ο μόνος τρόπος εφοδιασμού των εγκληματιών. Προφανώς όμως βλέπουμε ε, ότι πολλά ε, όπλα χρησιμοποιήθηκαν ε, για εγκληματικές δράσεις, τα οποία μάλιστα δυστυχώς απασχόλησαν με δραματικές συνέπειες στην επικαιρότητα. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε την νόμιμη και μη εγκληματική χρήση των όπλων. Είχα όμως ορισμένες ερωτήσεις προς τους παρεμβαίνοντες. σε ό,τι αφορά τις συλλογές και τα μουσεία πιο συγκεκριμένα. Θα μπορούσε να υπάρξει, μήπως είναι υπερβολική η εξαίρεση ε, από την οδηγία σε ό,τι αφορά τα παλαιά ε, όπλα, τις αντίκες. Μήπως είναι λοιπόν κάτι τέτοιο υπερβολικό. Γιατί ξέρουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε, για τέτοιους σκοπούς. Επομένω, εμένα μου φαίνεται ότι είναι μάλλον υπερβολικό το να τα εξαιρέσουμε εντελώ από την οδηγία. Και δεύτερον, για την συνελεσιμότητα, όπω ανέφερε και η Βίκη, εξεπλάγει όταν είδα ότι υπήρξε ε, ε αίτημα εξελασιμότητας με τη σήμανση μόνο των ουσιοδών μερών. Θα ήθελα όμως να ακούσω και τις δικές σα ε, απόψεις θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι γιατί εμένα μου φαίνεται μάλλον ε, περίεργο. Σέργιο Κοφεράτη, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας που μας δίνουν στοιχεία εξαιρετικής χρησιμότητας για τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Κάποιες σύντομες ερωτήσεις θέλω να θέσω για να μπορέσουμε κατόπιν να τις μετατρέψουμε σε νομοθετικό κείμενο. Συλλέκτες. Είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε ρητή εξαίρεση για ένα χωριστό κόσμο που είναι συλλέκτες. Τώρα, για τα μουσεία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, διαφορετικά από τα μουσεία για τους συλλέκτες, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες από χώρα σε χώρα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μία εξαίρεση για πράγματα που είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Πρέπει πρώτα να ενοποιήσουμε τους όρους που περιγράφουν αυτό το καθεστώς που θέλουμε να ρυθμίσουμε. Δεν ξέρω αν είναι δική μου δουλειά. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι. Ξέρω ότι είναι δική μου δουλειά αυτή, αλλά θα ήθελα να σα δείξω εσεί πώ βλέπετε να δώσουμε έναν ενιαίο χαρακτήρα σε κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Δεύτερον, πώληση online. Εξ αποστάσεως. Και εγώ αμφιβάλλω κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ένα κανόνα που να επιτρέπει την πώληση online. Μάλλον, να το πω αλλιώ πώληση online μπορεί να υπάρχει αν η χνηλασιμότητα και ο έλεγχος ε, των εμπλεκόμενων πλευρών εξασφαλίζεται. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μία, ένα πολλαπλασιασμό ανώμαλων καταστάσεων που ενισχύονται από ένα εργαλείο που μπορεί να ενθαρρύνει όχι μόνο την εμπορική δραστηριότητα αυτή καθ' αλλά και τον έλεγχο. Τέλος, εγκρίθηκε πριν από λίγο ο ελληνικός ε, ευρωπαϊκός κανονισμός για τις διαδικασίες απενεργοποίησης των όπλων. Δεν ξέρω αν λειτουργεί, δεν έχω καταλάβει αν αυτός ο κανονισμός λειτουργεί και ιδίω αν η, πραγματική, η απενεργοποίηση είναι πραγματική και κυρίω ε, αν άνευ επιστροφής, αλλιώς δεν θα υπάρχει πραγματική δυνατότητα ελέγχου. Αλλιώ μπορεί να έχουμε μια μορφή απενεργοποίηση που θα πρέπει να μπορεί πάντα να ελέγχεται από τις αρμόδιε αρχές. Αυτές είναι οι ερωτήσει μου. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που θα μου δώσετε. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Τοζίνσκι, μια παρατήρηση. Άκουσα κάποιους από τους Γάλλους ομιλητές χρησιμοποιούν τον όρο neutralize όταν μιλούν για deactivation. Το deactivate στα αγγλικά σημαίνει μόνιμα, χωρίς αναστροφή. Αυτό λένε οι Γάλλοι, πιστεύω, όταν χρησιμοποιούν τον όρο neutralized. Δηλαδή το, το, η εξουδετέρωση μπορεί να σημαίνει ότι απλά βγάζω ε, το βγάζω ότι αφαιρώ ένα κινητό ουσιώδες ε, στοιχείο. Καλύτερα να μιλάμε λοιπόν πάντα για απενεργοποίηση που σημαίνει ότι δεν μπορείς να αποκαταστήσεις την προτερή κατάσταση. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ γλωσσικά. Η αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πάντως να είμαστε σε μια τελική κατάσταση της εξουδετερωτήσης. Η Μάλη. Ευχαριστώ πρόεδρο. Με προλάβατε. Θέλω να επανέλθω στον όρο αυτό εξουδετερώνω, απενεργοποιώ για να τους ρωτήσω να μου εξηγήσουν αν έχει οριστικά χαρακτηριστικά ή όχι. Πάντως ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σας Στον κύριο Ήμπρη, συμφωνώ με όσα είπατε για, την, ε, για τα μουσεία και τους συλλέκτες. Νομίζω ότι τα όπλα, όπως ό,τι άλλο υπάρχει σε ένα μουσείο, πρέπει να μείνουν ως έχουν. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Και ένα δίδαγμα για το μέλλον. Για τους συλλέκτες, και εγώ θεωρώ πως η εθνική νομοθεσία αρκεί για την οργάνωση της δουλειά του συλλέκτη. Κύριε Σίλβης, έχω κάποιες ερωτήσεις μεταβραστικού χαρακτήρα. Δώστε κάποια νούμερα στο ξεκίνημα της παρέμβασής σας. Μπορείτε να τα ξαναδώσετε γιατί δεν είχα το χρόνο να τα σημειώσω. Λοιπόν, τάπα για την ε, απενεργοποίηση. Ο κύριος nobles. Ο ποτέ δεν μάλλον. Μιλήσατε για τις επιθέσεις ε, στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, τον Μερά για παράδειγμα, που είπατε ότι χρησιμοποίησε ένα παλιό όπλο του 1944. Εξεπλάγιν όταν ακούσαν, εξεπλάγιν ευνοϊκά όταν άκουσα να λέτε ότι υπάρχει δυσκολία κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην Ευρώπη. Έχετε κάποιες λεπτομέρειε, ας πούμε, ποια ήταν η ζωή αυτού του όπλου, που πού ερχόταν, πού το βρήκε τέλο πάντων. Έχετε κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Τέλος, προς όλους τους εμπειρογνώμονες. Έχετε αξιολογήσει το διαφυγόν κέρδος ή το συμπληρωματικό κόστος που θα επιφέρει η πρόταση επιτροπής σε όλους τους εμπλεκόμενους στο εμπόριο αυτό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. η Επιτροπή φαίνεται από τις ερωτήσεις ότι μοιάζει να έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που δεν έχει χαλάσει. Αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό ωστόσο είναι το εξής από την Επιτροπή. Πρώτον, μιλάμε για ημιαυτόματα που ομοιάζουν με αυτόματα. Πόσα είναι αυτά. Πόσα τέτοια όπλα υπάρχουν. Καταλαβαίνω ότι είναι μια αξιολογική ε, εικόνα, αλλά ποιος είναι ο ρυθμός. Γιατί αν θέλουμε να απαγορεύσουμε κάτι, καλό να ξέρουμε πόσα υπάρχουν. Δεύτερον, αν τα απαλωτριώσουμε, τα, τα, τα κατάσχουμε, κάπως πρέπει να αποζημιώσουμε τον κόσμο. Πόσο, ποια είναι η αξία τους, πόσο θα στοιχήσει. Αν τα πάρουμε και πληρώσουμε, τι αξία έχουν. Τελευταία παρατήρηση. Προσπάθησα να δω κάποιες στατιστικές για τον αριθμό των αδικημάτων που έγιναν με ε, νομίμως, ε, σε νόμιμη κατοχή τελούνται ή με αυτόματα όπλα. Υπάρχουν. Μπορεί να μου δώσετε ένα νούμερο. Ούτως ώστε να ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Διότι είναι πολύ δύσκολο να νομοθετούμε χωρίς αυτά τα βασικά δεδομένα. Ευχαριστώ. Thank you very much. So Ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα περάσω στην πρώτη ομάδα των τεσσάρων ομιλητών, όμως ε, πιστεύω ότι κάποιοι ίσως να θελήσουν να επανέλθουν σε αυτό το θέμα, όπως επίσης ε, και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν που θα κληθούν να μιλήσουν στο τέλος. Θα ήθελα να σας πω ότι η ε, αστυνομία της ε, των Βρυξελών αυτή τη στιγμή έκανε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. αυτό λέει. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να ε, συνεχιστεί η μάχη κατά της τρομοκρατίας και είναι σημαντικό αυτοί οι οποίοι διαθέτουν, οι νόμοι, οι πολίτες που τηρούν τους νόμους, αυτοί που διαθέτουν όπλα, ε, να εκπροσωπούνται και αυτοί. κάποιος ομιλητής που θα ήθελε να επιστρέψει ε, να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ κυρία Συγκεντρία. Το πρώτο στοιχείο για να σας δώσω ορισμένες διακρινήσεις ό,τι αφορά την απενεργοποίηση. Η απενεργοποίηση στη Γαλλία, ε, εξουδετέρωση, απενεργοποίηση είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι οριστική και μη αναστρέψιμη. Αυτό που σίγουρα θα αναφέρει και στη συνέχεια ο κ. Στασάν για την ε, απενεργοποίηση ή εξοδετέρωση. Δεν είναι ποτέ τέλεια αυτή η διαδικασία. Προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο ε, συγκεκριμένοι και εντελεχεί, όμω πάντα βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψει και προσπαθούμε να τι διορθώσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Γαλλία μετά από όλε αυτέ τι δολοφονίε, ότι προσπαθούμε ε, να βελτιώσουμε την ανταπόκρισή μα. Ο ισχύων κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξάλλου, προβλέπει ακριβώ μία διαδικασία διόρθωση. Αυτό για την επανεργοποίηση, για την ειχνηλασιμότητα. Έχουν αναφερθεί πολλέ ερωτήσει. Προφανώ η ειχνηλασιμότητα για τι αστυνομικέ αρχέ είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γιατί πάντα αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες έτσι καλώ τα όπλα, τα στρατιωτικά τα λεγόμενα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη ε, οδηγία και έτσι είναι δύσκολο να, τις ε, ανοιχνεύσουμε, να τα ανοιχνεύσουμε. Παρότι στην αρχή ήταν νόμιμα ε, και στη συνέχεια κάπως εξαφανίστηκαν από, τον, από την νόμιμη αγορά και είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε. Πάντα λοιπόν υπάρχει αυτό το ζήτημα της εθελεσιμότητας. Μετά, μάλλον εγώ δεν το ανέφερα αρκετά σαφώ, αλλά είναι δύσκολο το ζήτημα. Για την συνδεσιμότητα λοιπόν, από την αναθεωρήση τη οδηγία 2008, έχουμε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε σε εθνικό επίπεδο για την χνηλεσιμότητα στο πλαίσιο τη χώρα. Το πρόβλημα είναι στι ενδοευρωπαϊκέ μεταφορέ. Όταν ένα όπλο το αγοράζει κάποιο που ταξιδεύει για να αγοράσει ένα όπλο ή το παραγγέλνει από το εξωτερικό. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των εθνικών μητρώων και αρχείων, κάτι το οποίο είναι δύσκολο βέβαια να εφαρμοστεί, εφόσον ο καθένας έχει φτιάξει τα δικά του μητρά με τους δικούς του ε, κανόνες. Έχουμε λοιπόν κάποιον που πάει από τη μια χώρα στην άλλη για να αγοράσει το όπλο. Και η διαδικασία αυτή τη στιγμή για την ενδοευρωπαϊκή αυτή μεταφορά γίνεται με συγκεκριμένα έγγραφα. Υπάρχει άδεια που πρώτα εκδίδεται από τη χώρα που χορηγεί αυτή την άδεια και μετά έχουμε και μια άδεια μεταφοράς από τη χώρα στην οποία γίνεται η αγορά του ε, προϊόντος. Όμως είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο έχει και την ε, άδεια και το έγγραφο αυτό. Επομένω δεν ξέρουμε ποιο είναι το όπλο ακριβώς που αγόρασε και θα μεταφέρει, ούτε πότε θα γίνει η αγοραπολισιακή μεταφορά και δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των δύο εθνικών αρχείων και μητρών. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κενό στην εκνελεσιμότητα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Αυτό θέλουμε να διορθώσουμε. Και μάλιστα είναι ένα ζήτημα το οποίο υπήρχε και μετά τις επιθέσεις στο Λονδίνο και στη Μαδρίτη για τις εκρηκτικές ύλες. Ο κύριος Ιμπέη. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια σειρά ερωτημάτων όσον αφορά τη σχέση ε, συλλεκτών ε, και τα μουσεία. Και νομίζω ότι το βασικό είναι ε, να πούμε ότι αυτό για το οποίο μιλάμε, για το αντικείμενο που μιλάμε, ασχέτως του ποιος το κατέχει, πρόκειται για πολιτισμική κληρονομιά. Οι ε, συλλογέ αποτελούνται, ε, ανήκουν κυρίως ε, σε ιδιωτικούς συλλέκτες και έτσι περιορίζουμε την πρόσβαση στο κοινό σε περίπτωση που αυξηθούν αυτές οι ε, συλλογές. Τώρα όσον αφορά την ασφάλεια των μουσείων έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου έχουν κλαπεί ε, αντικείμενα από μουσεία όμως δεν έχουμε υπόψη μα περιπτώσεις που έγινε για να χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Μιλώ για την Αγγλία, για την Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύουμε πως ναι ισχύει δεν πουλούμε όπλα της συλλογή μας, δεν μπορείτε να πάρετε κάποια όπλα από τη δική μας συλλογή. Ε, η ασφάλεια μας είναι πάρα πολύ αυστηρή, υπάρχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση και έχουμε ένα καλά σχεδιασμένο ε, σύστημα ασφαλείας Υπάρχει ε, πρόσβαση για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όμως ε, ε, ελέγχονται εκτενώς ούτως ώστε να έχουν έναν καλό λόγο για τον οποίο βρίσκονται εκεί. Καταγράφουμε ποιοι έρχονται, τους εξετάζουμε όταν καταφθάνουν Και το βασικότερο, όταν αποκτούμε κάτι, τότε ακολουθούμε όλη την νόμιμη διαδικασία για να, να βεβαιωθούμε από πού προήλθε ε, και να μάθουμε όλη την ιστορία του. Η ασφάλεια των ιδιωτικών ε, συλλογών στην ε, Αγγλία. Τα όπλα εκεί κατηγορίας Α ήταν παράνομα, είναι παράνομα εδώ και αρκετό καιρό, όμως η άδεια για τα όπλα είναι πάρα πολύ αυστηρή στην Αγγλία και νομίζω ότι είναι αρκετά καλή για το σκοπό που εξετάζουμε. Τώρα, ε, για το αν θα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση για τα μουσεία από την οδηγία, αν κάτι τέτοιο είναι υπερβολικό, εγώ δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό, διότι η εξαίρεση δεν θα εξαιρέσει τα μουσεία από το να κάνουν τους αυτηρούς ελέγχους που ήδη κάνουν τα μουσεία έχουν αυστηρή ε, νομοθεσία ε, και αυτό ισχύει ιδιαίτερως για το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να είμαι ε, ειλικρινής για αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει επαρκής προστασία. Οι συλλέκτες και σχετικά με το άμα είναι χαλαρός ο ορισμός υπάρχουν διάφοροι ορισμοί σχετικά με το τι είναι συλλέκτης και τώρα θα ήθελα να προτείνω μερικούς από αυτούς που βοηθούν όμως αυτό που συστήνω όσον αφορά την απάντηση σε ένα ερώτημα είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μονάχα μια κοινή, ένα κοινό όρο σχετικά με το τι είναι ένα συλλέξη στην Ευρώπη, αλλά και εναρμονισμένες συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορεί κανείς να επιτρέπεται ε, να έχει ένα όπλο και να το αποθηκεύει βέβαια. Ένα τελικό ερώτημα σχετικά με το κόστος της επενεργοποίησης. Ναι, εμείς το μουσείο το εξετάσαμε, όπως επίσης ε, και το Αυτοκρατορικό Μουσείο και υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περί το 1 εκατομμύριο λίρες να απενεργοποιήσουμε κάθε συλλογή. Δεν αξίζει διότι ποτέ δεν θα, τα δεν θα το πουλήσουμε όμως το κόστος για την καταστροφή τους ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια λίρες. Ο κύριος Ευχαριστώ. Πρώτον, η σήμανση των ουσιοδών ε, συστατικών. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, η οδηγία προβλέπει ότι η σήμανση πρέπει να είναι ε, σταμπαρισμένη σε ένα ουσιώδες ε, συστατικό στοιχείο του συναρμολογημένου όπλου. Αν υπάρξει, υπάρχει ένα δεύτερο εδάφιο που λέει ότι όλα τα ουσιώδη ανταναρκτικά που πολλούνται πρέπει να, είναι, να έχουν σήμανση και άδεια για τον πολιτή. Αυτό σημαίνει ότι αν η καταστροφή ενός ουσιώδου συστατικού του συναρμολογημένου πυροβόλου καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο ουσιώδες ε, στοιχείο που επίσης έχει σήμανση και χρειάζεται άδεια για να το λάβεις. Υπάρχει λοιπόν μία συμμόρφωση για να μην υπάρχουν ανταλλακτικά που δεν έχουν σήμανση αφενός και αφετέρου αποφεύγουμε τη γραφειοκρατία έχοντας ε, πολλούς αριθμούς στο ίδιο όπλο. Επιπλέον, η πρόταση της Κομισιόν είναι σωστή γιατί προτείνουν να γίνει ομοιόμορφο το σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε κάθε κατασκευαστής που και κάθε εισαγωγέας όπλων να έχουν ε, σήμανση του ίδιου προϊόντος, του ίδιου συστατικού, ούτω ώστε να μην έχει το ενδεχόμενο ε, αλλού σε μια χώρα να, να βάζει τη σήμανση στην Κάνη, αλλού να βάζει στην ε, Σκανδάλη, αλλού και έτσι να μην έχει τα συστατικά, ε, τα ουσιώδη συστατικά ίδια παντού, άμα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ανταλλακτικό. Δεν ξέρω, είναι σαφέστερα αυτά που λέω. Ναι, δεν ξέρω πόσο εφικτά είναι, αλλά είστε σαφείς. Ο κύριος Πότεβε. Έχω κι άλλες απαντήσεις να δώσω. Με συγχωρείτε. Κοράτσα Μπίλτ ζήτησε κάποια παραδείγματα για το τι νομίζουμε για την ομοιομορφία της νομοθεσίας ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Εμείς νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το σύστημα ομοιόμορφο σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Για παράδειγμα, η Επιτροπή είχε τη δυνατότητα να επαληθεύσει ότι σε κάποιες χώρες η οδηγία εφαρμόζεται με τον α τρόπο, σε άλλες με άλλο. Κατά συνέπεια είναι χρήσιμο να κάνει το σύστημα ομοιόμορφο για να αποφύγεις αυτές τις, ε, ε, αυτέ, αυτά, τα, αυτές τις τρύπες. Τώρα, για την απενεργοποίηση. Η απενεργοποίηση ήδη έχει γίνει σωστά. Κάποιες χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία το έχουν πετύχει. όχι με τον ίδιο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο όμως επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό είναι αν υπάρχει πιστοποιητικό. Αυτό το όπλο είναι καλά, είναι απενεργοποιημένο, θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα πιστοποίησης μιας ε, απενεργοποίησης. Για παράδειγμα, για τα όπλα συναγερμού σηματοδότηση στην Ιταλία και τη Γερμανία εδώ και 10 χρόνια. Ήδη παράγουμε όπλα συναγερμού σηματοδότηση που δεν μπορούν να μετατραπούν. Αν μετατραπούν, ε, έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν επιτρέπουν την μετατροπή τους. και δεν μπορεί να τα χειριστείς με σωστό τρόπο όπλα που έχουν φτιαχτεί για σηματοδότηση. Και ο κύριος Κοφεράτη έθεσε μια ερώτηση για την απενεργοποίηση. Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε ένα όργανο πιστοποίησης που θα λέει ότι η απενεργοποίηση έγινε σωστά και το απενεργοποιημένο όπλο είναι ασφαλές. να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή. Μαλίν, τα στοιχεία είναι όλα στη στην ε, ιστοσελίδα. Όλες αυτές οι παρουσιάσεις είναι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. Έχουμε μισή ώρα καθυστέρηση σχεδόν. Ζαλουίκ Στάσεν. Oh, oh um, Α, ναι, συγγνώμη, ο κύριος Πατεβά ήθελε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εν συντομία, πολλά ακούστηκαν κυρίως να στο διαδίκτυο, τους διαμεσολαβητές, πρέπει να έχουμε κατά νου για τους ενδιαμέσους συμμεσάζοντες. Ε, Διακύβημα εδώ είναι ε, η καλύτερη στεγανοποίηση μεταξύ της νόμιμης και παράνομης σφαίρας. Όπως ε, αναφέρθηκε προηγουμένως, πλέον βλέπουμε ότι όσοι θέλουν να εγκληματίσουν στρέφονται προς παλαιά όπλα ή απενεργοποιημένα όπλα, τα οποία ενεργοποιούν στη συνέχεια εκ νέου. Γιατί υπάρχουν ένα, υπάρχει ένα πολύ καλό σύστημα ελέγχου στην Ευρώπη, παρά τις ε, όποιες δυσκολίες, όμως βλέπουμε ότι είναι κάτι το θετικό τουλάχιστον, ότι εκεί έγκυται το πρόβλημα και έχει αλλού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, να εξετάσουμε, να εντοπίσουμε ε, τυχόν ελλείψεις και κενά στην ομοθεσία και τώρα και να δούμε τι θα έχει γίνει όταν θα εφαρμοστεί η οδηγία. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει δυνατότητα εναρμόνιση του καθεστώτος των συλλεκτών που δεν έχει γίνει ακόμα στην Ευρώπη και να θέσουμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ε, μπορεί να διαμορφωθεί μια συλλογή. Είναι σημαντικό να καλύψουμε πλήρως το θέμα του διαδικτύου και σε ό,τι φορά την πρόταση της οδηγίας που έχει ως στόχο να περιορίσει τις πωλήσει στο διαδίκτυο, αυτό να συμπληρωθεί και με τις αγορές στο διαδίκτυο. Και η πόλη, λοιπόν και η αγορά στο διαδίκτυο είναι σημαντικό στοιχείο γιατί ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφέρει η νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών και έτσι μπορούν κάποια ε, όπλα, ε, να μην υπάρχουν πλέον στην, χώρα Α, αλλά με μεγάλη ευκολία να μπορεί να τα βρει κάποιο στη χώρα Β. Και νομίζω ότι με αυτό το πνεύμα θέλησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, υποβάλει την πρόταση και για το θέμα του διαδικτύου. Και για τα μουσεία. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό ε, που γίνεται στην Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει σε όλα τα κρατημέλη. Να, υπάρχουν λοιπόν κοινοί όροι σε ό,τι αφορά ε, τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τα μουσεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επόμενος ομιλητής, ο Ζων Λουίξ Τασάν από το Βέλγιο, είναι υπεύθυνο ελέγχου όπλων. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο ως διευθυντής ε, του, ε, της του αρμόδιου φορέα ελέγχου των ε, όπλων. Προτίμασα την παρουσίασή μου μαζί με τη συνάδελφο Δέξου Αριστερών από, τις, από την υπηρεσία ελέγχου της διακίνησης όπλων. Θα ήθελα να της δώσω το λόγο για πολύ λίγο. Είναι σημαντικό το ζήτημα το οποίο εξετάζεται σήμερα, αλλά και ποια είναι τα ουσιώδη συστατικά μέρη, ε, ποιο είναι το όπλο συναγερμού. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, 4-5 χιλιόμετρα από εδώ, έχουν υπάρξει πυροβολισμοί, τρεις αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, σε απόσταση 5 χιλιόμετρων τρει αστυνομικοι εχουν τραυματιστει σε εδώ. Και αυτό το όπλο το οποίο αναφέρεται από τον τύπο ως Καλάσνικοφ ε, θα πρέπει να δούμε από πού έχει προέλθει, και γι' αυτό είναι και σημαντική, αποδεικνύεται ότι είναι σημαντική η Να δούμε ποια είναι τα ουσιώδη μέρη. Αν είναι ένα όπλο το οποίο προήλθε από, από μια ιδιωτική συλλογή. Αν είναι ακουστικό που έχει μετατραπεί. Όλα αυτά απαιτούν μια εναρμόνιση. Αυτή τη στιγμή οι τρεις ε, τραυματίες ε, αστυνομικοί ευτυχώς δεν είναι ε, άμαχοι. Πρέπει να, να το εξετάσουμε περαιτέρω. Όλα αυτά όμως αποδεικνύουν τη σημασία ε, και πόσο επίκαιρο είναι και αυτό το θέμα που εξετάζουμε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, θα αναφερθώ στα ημιαυτόματα, τα άσφαιρα και την απενεργοποίηση των όπλων. Και επανέρχομαι σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Το disactivation στα αγγλικά είναι το neutralisation στα γαλλικά. Το ίδιο πράγμα σημαίνει απενεργοποίηση. Είναι λοιπόν επιμέρους ε, διαδικασίες που ακολουθούνται, ούτω ώστε να μην μπορεί κάποιος να ε, πυροβολήσει με αυτό το όπλο. Και αυτό είναι μάλιστα μια αναστρέψιμη διαδικασία. Πρέπει να μιλήσουμε για το καθεστώς των ε, συλλεκτών και πρέπει οπωσδήποτε να προβλέψουμε και να προσδιορίσουμε το ειδικό καθεστώς του συλλέκτη. Υπάρχει ήδη αυτό το καθεστώς με μεγάλη επιτυχία σε ορισμένε χώρες το καθεστώς του συλλέκτη θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει τους ιδιωτικούς, τους ιδιώτες ε, συλλέκτες, ε, τα, τα μουσεία δημοσίου δικαίου και τα μουσεία ιδιωτικού δικαίου. Πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε αυτό το καθεστώς στο πεδίο εφαρμογή ε, της οδηγίας και να δώσουμε τη δυνατότητα συλλογή όπλων κατηγορίας Α για αυτούς τους συλλέκτες, οι οποίοι βέβαια έχουν την απαραίτητη άδεια οι προποθέσει, οι όροι παράδοση και χορήγηση μάλλον αυτή τη άδεια για του συλλέκτε όπλων θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα ο περιορισμό τη συλλογή ε, σε συγκεκριμένο ε, διάστημα 20 χρόνια ε, κατά μέγιστον. Δεύτερο, περιορισμός του συνολικού αριθμού των όπλων που μπορεί να συλλέξει κάποιος. Ίσως θα μπορούσαμε εδώ να δούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ιδιωτικού συλλέκτη, ε, του ιδιωτικού μουσείου ή του δημοσίου μουσείου. Μετά, ε, ε, περιορισμός του συνολικού αριθμού των αυτομάτων όπλων που συλλέγονται κατά μάρκα και κατηγορία. Γνωρίζω ότι μπορεί να υπάρξουν και πάλι διαφορές μεταξύ των τριών κατηγοριών που προανέφερα. Και τέλος, επιβολή ε, προϋποθέσεων αποθήκευσης με πιο συγκεκριμένους κανόνες για την αποθήκευση αυτόματων όπλων με την απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιώδων μερών, που είναι ουσιώδη δηλαδή για την ε, χρήση του όπλου. Τώρα περνώ στο ζήτημα ε, το οποίο μου ζητήσατε να παρουσιάσω, τις κατηγορίες όπλων. Εδώ λοιπόν μιλήσαμε για την απενεργοποίηση των όπλων. Απενεργοποιημένο λοιπόν όπλο, αυτόματα ή όχι. Σκοπός της απενεργοποίησης, όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι να καταστήσουμε τα όπλα και μάλιστα με, με μια αναθέσιμη διαδικασία, να, ώστε να μην είναι πλέον σε θέση να πυροβολήσει κάποιο με αυτά. Από τις 8 Απριλίου 2016 και μετά υπάρχουν ε, για τα όπλα που υπάρχουν ήδη χωρίς ε, μεταπόλησή τους δεν υπάρχει τροποποίηση. Και τροποποίηση θα υπάρξουν μόνο αν υπάρξει και μεταπόλησή τους. Λοιπόν, η παράδοση, χορήγηση ενός πιστοποιητικού μιας άδεια θα ισχύει για τα 28 κρατη Βάσει τις οδηγίες 91 477 Αυτά τα απενεργοποιημένα όπλα, είτε είναι αυτόματα είτε όχι, δεν συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναγκαιότητα όμως η χνηλαστιμότητα των όπλων αυτών παραμένει και έτσι απαιτεί την ταξινόμηση αυτών των όπλων τουλάχιστον στην κατηγορία Δ, αλλά ε, το ιδανικό θα ήταν να μπουν στην κατηγορία Γ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη αυτόματα όπλα ε, μη στρατιωτικού τύπου που μοιάζουν με αυτόματα. Ε, χρησιμοποιείται λοιπόν το civilian έναντι του στρατιωτικού. Πρόκειται λοιπόν για μακρύκανα ε, μη στρατιωτικά ή μη αυτόματα ε, όπλα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μοιάζουν λοιπόν με αυτόματα, αλλά αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και υποκειμενικό αν θέλετε. Και έτσι θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ των μελών. Αυτό το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί στο Βέλγιο και το έχουμε καταλήψει γιατί είδαμε ότι ήταν ανεφάρμοστο. Αυτό το υποκειμενικό κριτήριο θα οδηγήσει σε σύγχυση και σε χάος μέσα σε μερικά χρόνια. αυτό το χάος που θα δημιουργηθεί μεταξύ των εθνικών ερμηνειών ε, θα ευνοήσει σίγουρα μόνο το εγκληματικό, τα εγκληματικά κυκλώματα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Θα ήταν σκόπιμο να νομοθετήσουμε ενδεχομένω σε, ό,τι αφορά τις θήκες ε, και να έχουμε την ίδια ταξινόμηση ε, με το όπλο ε, για το οποίο χρησιμοποιείται. Και αυτό το όπλο μπορεί να αποτελέσει ουσιώδες μέρος του όπλου. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει νοσημότητα και εδώ. Για παράδειγμα, σε μία ημιαυτόματη καραμπίνα μπορούμε να περάσουμε από τις, από τις 30 στις 10 θήκες. Επομένως, περιορίζεται πλέον ε, ο αριθμός ε, των θήκων που μπορούμε να έχουμε. Επιπλέον, θα πρέπει οι θήκες αυτές πρώτον να ακολουθούν την κατηγορία όπλου για την οποία χρησιμοποιούνται, να, έχουν, να περιοριστεί ο αριθμός ε, και να ταξινομούνται πλέον ως ουσιώδη μέρη του όπλου που υπάρχονται έτσι και στους κανόνες της μελασιμότητας δηλαδή ε, αδειοδότηση της διατήρησης ε, ε, αριθμού σειράς και χνηλασιμότητα. Τα αυτόματα που έχουν μετατραπεί σε αυτόματα. Προτείνουμε τη διατήρηση της αξινόμησης αυτών των όπλων στην κατηγορία Β. Αρκεί η μετατροπή να έχει πραγματοποιηθεί από δημόσιες ιδιωτικές αρχές ή από εξουδετημένα πρόσωπα βάσει και της εθνικής νομοθεσίας μέσω μιας διαδικασίας που διασφαλίζει το μη αναστρέψιμο της μετατροπής. Παίρνουμε λοιπόν στη διαδικασία της ε, απενεργοποίησης με Συγκεκριμένε ε, διατάξεις, προποθέσει και ένα πιστοποιητικό το οποίο να μην μπορεί ε, να παραποιηθεί. Για τα πυροβόλα όπλα, μάλλον συγγνώμη, ε, του συναγερμού, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των αρχικών όπλων συναγερμού και των όπλων συναγερμού που τα οποία έχουν μετατραπεί σε όπλα συναγερμού. Για την πρώτη κατηγορία, είναι όπλα τα οποία δεν έχουν σκοπό αρχικά ε, να έχουν ουσιαστικά φυσίγγια μέσα. Είναι κρότου μόνο. Διαμορφώθηκε λοιπόν μία ομάδα εργασίας κατόπιν ετήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσδιορίσουμε ακριβώς ενιαία τεχνικά κριτήρια. Διακόπτη Πρόεδρος, λυπάμαι πάρα πολύ. Μπορείτε ε, να συντομεύετε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μισό λεπτό. Για τα μετατρέψιμα όπλα συναγερμού, ακουστικά και κρότου δηλαδή, που χρησιμοποιούνται για παραστάσεις, ο ορισμός τους είναι με τα μετατραπέντα πραγματικά όπλα για να ρίχνουν ε, άσφαιρα πυρά. Η διαδικασία πρέπει να ε, παρακολουθείτε και δεν μπορεί να αφήνεται στην, ε, στην ελεύθερη επιλογή του ατόμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στραφεί στην διαδικασία μετατροπής των όπλων αυτών που πρέπει να παραμείνουν να υπάγονται στην αρχική τους κατηγορία και οι επιχειρήσεις που τα θέτουν στη διάθεση ε, άλλων για διαφορετικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν τις αναγκαίες και απαιτούμενες άδειες. Τώρα, ο, απο, απομιμήσεις όπλων, όπλα δηλαδή που μοιάζουν με τα πραγματικά και χρησιμοποιούν ε, ε, καύση, ε, σύστημα εσωτερικής καύσης για την εκπομπή ε, σφαιρών, άσφαιρων σφαιρών. Πρέπει να αλλάξει η οδηγία στο σημείο αυτό προβλέποντας να υπάρχει να περιγράφονται ως πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και ε, ε, συστατικά, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν και τον σιγαστήρα και την ε, θήκη. Στην κατηγορία Β, που αυτά τα όπλα που υπάγονται σε νομοθεσία συμπεριλαμβανομένης και της θήκης, ενώ η Γ είναι τα όπλα που υπάγονται σε δήλωση και μια κατηγορία δέλτα που είναι τα υπόλοιπα όπλα. Τελειώνω, τελειώνω. Ο ορισμός των ουσιοδών συστατικών. Μιλάμε για το θέμα αυτό επιμακρό. Εγώ κάνω μια πρόταση που βασίζεται στην απόφαση και την νομοθεσία του CIP. Όπλα αυτόματα ή μη αυτόματα, όπως κάθε στοιχείο μεταξύ κάνει ε, ε, και μυστήρας διακόπτει ο πρόεδρος. Μπορείτε να μας στείλετε γραπτός. Γραπτός μπορείτε. Ωραία, χωρίς πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Φίλιππο Σεγκάτα. Από την Ένωση Κυνηγών της Ένωσης. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Ανά. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Κυνηγών και Συντήρησης της Φύσης στην Ένωση. Υπάρχουμε από το 1977, στις Βρυξέλλες εδρεύουμε, εκπροσωπούμε 7 εκατομμύρια κυνηγούς. Είμαστε οι μεγαλύτεροι εμπλεκόμενοι φορείς στις συζητήσεις. Έγινε πολλής λόγος για την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα, εγώ θα αλλάξω το πλαίσιο. Τι είναι το κυνήγι σήμερα, τι κάνουν οι κυνηγοί και γιατί χρειάζονται όπλα. 16 δις τζίρο έχει το κυνήγι στην Ευρώπη. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης ε, της ε, φύσης και της προστασίας των οικοτόπων. Είναι μια υπηρεσία οικοσυστήματος που βοηθάει την αγροτική οικονομία, μακρά παράδοση ριζωμένη στην κουλτούρα της Ευρώπης και μια βιώσιμη πηγή υγιεινής διατροφής. Μην το ξεχνάτε. Βγαίνει ο κυνηγό, φέρνει κυνήγι στο σπίτι. Αυξάνεται η δημοφιλία του κυνηγιού σε κάποιες χώρες για, το, για τα τρόφιμα, για την τροφή δηλαδή. Στην Σουηδία για παράδειγμα το 87% του πληθυσμού εγκρίνει το κυνήγι και όλο και περισσότερες γυναίκες κυνηγάνε και ζητάνε άδειες για να αποκτήσουν μια εμπειρία της φύσης. Η θέση μα για την πρόταση τώρα. Καλωσορίζουμε την αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη Δημοκρατίας. Αυτό είναι σαφέ. Πρέπει να είναι σαφέ. Υποστηρίζουμε του σωστού ελέγχου των όπλων και τις δικαιολογημένες, ε, και τους δικαιολογημένους και αναλογικούς περιορισμούς στην αγορά και κατοχή. Τα μέτρα που συζητούμε λοιπόν για τη σήμανση, την ανιχνευσιμότητα, την διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών είναι πρόσδεκτα. Όπως και άλλοι ομιλητές, σημειώνουμε ότι η Επιτροπή δεν συνόδευσε την πρόταση τροποποίηση με μελέτη αντικτύπου. Φοβόμαστε ότι τα μέτρα που προτείνονται μπορεί να έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στην νόμιμη χρήση των όπλων. Ήδη έχουμε υποβάλει μέχρι του ESSF που είναι η κοινή μας οργάνωση μια κοινή θέση που απαντάμε στο έγγραφο εργασίας προτείνοντας λύση επαναλαμβάνουμε, Συχνά τονίσαμε ότι η πρόταση αυτή ε, δεν μπορεί να περιλαμβάνει ε, ζητήματα που είναι άσχετα με τα όπλα όπως οι, ποιοι είναι οι νόμιμοι χρήστες. Εμείς πάντα είπαμε, η Επιτροπή μάλλον είπε ότι ο στόχος της πρότασης δεν έπρεπε να είναι η κυνηγή. Φοβόμαστε ωστόσο ότι θα υπάρχει μια δυσανάλογη επίπτωση σε εμά. Θέλουμε να αλλάξουν λοιπόν αυτές οι προτάσεις ε, που έχουν σαν έμεση επίπτωση να πλήξουν τους κυνηγούς. Αυτό είναι ένα καλάσνικο, δεν χρησιμοποιείται για για απαγορεύεται. Είναι ε, κατηγορία Α. Εμεί δεν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό. Έχουμε όμω αυτά. Άλλ, έχουμε όπλα κυνηγιού σε άλλε κατηγορίε. Ε, στα ε, μακρύκανα, στα ημιαυτόματα κοντόκανα, περίστροφα, ε, μα, ε, όπλα δίκανα και άλλα τέτοια όπλα που ανήκουν στις κυνηγιού που ανήκουν στην κατηγορία. Επίσης και στην κατηγορία Δέλτα έχουμε τα μονόκανα, τα μακρύκανα με, διπλή, ε, με διπλό γεμιστήρα κτλ. Τώρα, για τα β το πρόβλημα προκύπτει από αυτό το ημιαυτόματο που είναι για μη στρατιωτική χρήση που μοιάζει όμως με όπλο αυτό με, αυτό με το μηχανισμό. Όλοι το λένε αυτό το, το αναφέρουν αυτό το όπλο, αλλά αυτό καθ' αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα δημοφιλές όπλο κυνηγιού. You... Oh, not working very well. Θέλω να σας δείξω το πρόβλημα που έχουμε. Βλέπετε εδώ, σύμφωνα με την πρόταση, αυτό το ημιαυτόματο όπλο που μοιάζει με αυτόματο θα τεθεί στην κατηγορία, θα υπαρχθεί στην κατηγορία Α, λόγω της ομοιότητάς του. Αισθητικά, της αισθητικής παρουσίασής του. Τι θα γίνει όμως μετά. Στην κατηγορία Α θα έχουμε έναν ημιαυτόματο μηχανισμό που θα μοιάζει με όπλα της κατηγορίας Β. Άρα θα υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ απαγορευμένου ημιαυτόματου και μη απαγορευμένου όπλου και μας ανησυχεί τι θα γίνει στο μέλλον για αυτά τα ε, ε, πυροβόλα όπλα. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή μοιάζουν με κάτι απαγορευμένο, να μπουν και αυτά σιγά σιγά στην κατηγορία των απαγορευμένων και να φύγουν από την ομάδα των ε, κυνηγετικών όπλων. Εγώ σας προσπαθώ να σας εξηγήσω γιατί υποστηρίζουμε την κατηγορία αυτή. Έχουμε μια πρόταση. Εφόσον η Επιτροπή δηλώνει ότι το παραγματικό πρόβλημα προκύπτει από τη μετατροπή των αυτόματων όπλων σε ήμι αυτόματα, και αυτό είναι ο λόγος τον οποίο η κατηγορία αυτή αρχικά είχε δημιουργηθεί, προτείνουμε να εισάγουμε κοινά πρότυπα μετατροπής που εξασφαλίζουν κάθε μετατροπή πυροβόλου όπλου που αλλάζει την κατηγορία του να γίνεται με τρόπο που θα καθιστά την μετατροπή αυτή μη αναστρέψιμη. Περίπου αυτό που πρότεινε ο κ. Στάσενς πριν λίγο. Ενιαία, ομοιόμορφη λύση. Να εμποδίσουμε δηλαδή το να μετατραπούν σε πλήρως αυτόματα τα όπλα αυτά ξανά. Η οργάνωσή μου πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα να μπει στην ε, οδηγία μια ρύθμιση όπως αυτή που σας περιέγραψα. Επίσης έχουμε και μια παρατηρήση για τις πωλήσει online. Έγιναν πολλές συζητήσει για το θέμα αυτό. Βάσει της οδηγίας για τα μέσα Επικοινωνία εξ η πώληση online δεν απαιτεί ταυτόχρονη φυσική παρουσία. Η φυσική παρουσία λοιπόν έχετε σε αντίθεση με το γράμμα της οδηγία. Επίσης μας φοβίζουν άλλα χαρακτηριστικά της εξαποστάσεως πώληση, όπως τα email, τα τηλέφωνα, οι συζητήσεις στο τηλέφωνο που όταν γίνει εθνική ενσωμάτωση μπορεί να μετατραπούν σε εγκληματικό, σε εγκληματική δράση. Αυτά. Τελειώνω, πρόεδρε. Όπως είπε και ο κ. Σκοφεράτη, η οργάνωσή μου υποστηρίζει τον αυστηρό έλεγχο από τις αρχές των πωλήσεων με ίντερνετ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανιχνεσιμότητα στην ε, ειρήνη. Η έμφαση στην οδηγία θα πρέπει να είναι το σκοτεινό δίκτυο, όχι η νόμιμη πώληση online. Ζητούμε λοιπόν από το Κοινοβούλιο να αποφύγει την διάκριση μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων χρηστών όταν εξετάζουν την νόμιμη πώληση, τη νόμιμη χρήση των πωλήσεων online. Προτείνουμε λοιπόν να επανέλθουμε στην αρχική νομοθεσία. Οι σιγαστήρες, τα μηχανήματα μείωσης του ήχου, θεωρείται ότι δεν, υπόθηκε ότι δεν δημιουργούν κίνδυνο στην ασφάλεια. Και για την οδηγία αυτή οι σιγαστήρες δεν θα έπρεπε να θεωρούνται ως ουσιώδες στοιχείο. 20 δευτερόλεπτα. αποθήκευση. Ε, συζητείται όλο και περισσότερο. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν υπάρξει μια ρύθμιση για την ασφαλή αποθήκευση των όπλων και κατηγοριών Α και Β και να αποφεύγουν τρόπους πιθανότητα πρόσβασης από άτομα χωρίς άδεια. Τα κράτη-μέλη όμως θα πρέπει να βρουν τον καταλληλότερο τρόπο ρύθμισης του θέματος της αποθήκευσης. Άλλες προτεραιότητες θα πρέπει να υπαχθούν όπως και τώρα στην αρχή της επικουρικότητας και να αφήσουμε στην εθνική νομοθεσία το πότε θα δίνει και θα φερεί τις άδειε. Συμπεράσματα πρόεδρε, τα είπαμε. Ευχαριστώ. Ε, δεν κόβω 18, 7 εκατομμύρια κυνηγούς, να αυξηθούν ωραία, αλλά πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο και στα μέλη και στους υπόλοιπους ομιλητές. Θα δώσω το λόγο στο Stockholm Peace Research Institute και στη Europol. Και μετά, αν έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Εντάξει. να πάει σε μια ψηφοφορία η εκπρόσωπο της Λίβεο που θα προέδρευε αυτή της ε, συνεδρίασης. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να περικόψω πάρα πολύ ε, την ε, παρουσίασή μου για να μην επαναλάβω πράγματα τα οποία έχουν ήδη υποθεί. Όσον αφορά ε, την Σύπρη, ε, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα πιο ολιστικά, ούτως ώστε να, αναλάβουμε, να αναφερθούμε στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ε, οι αρχές ασφαλείας, αλλά και οι πολίτες. Η πρόσβαση σε όπλα και τρομοκρατικές δραστηριότητες είναι μονάχα ένα κομμάτι. Όταν μιλάμε με την κοινότητα των υπηρεσιών ασφαλείας, μιλούμε την αύξηση παρατηρείται μια αύξηση των όπλων ενώ αρκετά κράτη-μέλη έχουν κάνει έρευνες και δείχνουν ότι ε, τα ποσοστά ε, χρήσης όπλων ε, σε δολοφονίες έχουν μειωθεί σε σχέση με άλλα, άλλες περιπτώσεις. Ε, πολλοί δέχονται ε, κάποιες αλλαγές ε, σε αυτό το θέμα και βλέπετε ότι το ζήτημα αυτό ε, καλύπτει ένα μεγαλύτερο εύρο όπλων όπως είναι για παράδειγμα τα ημιαυτώματα στα οποία επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερως. Κάτι για τα ημιαυτώματα διότι διότι πολλή έμφαση δίνεται σχετικά με την μετατρεψιμότητά τους και εμείς δεν έχουμε πιστεί ότι αυτό είναι το μοναδικό ζήτημα ασφάλειας το οποίο σχετίζεται με τα ημιαυτόματα όπλα θα πρέπει να απομονώσουμε τα χαρακτηριστικά των ημιοαυτόματων όπλων, ούτω ώστε να μην γίνονται ελκυστικά στου ε, εγκληματίε, διότι ακόμα και αν υπήρχε διαθεσιμότητα ημιοαυτόματων όπλων, ε, σε όπλα τότε τα ημιοαυτόματα ήταν αυτά τα οποία θα επέλεγαν, διότι ε, ο έλεγχο των βολών έχει ω αποτέλεσμα να μπορούν να μην ξοδεύουν πολλέ σφαίρε, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν ανεξέλεγκτου στόχου. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε την ελκυστικότητά τους στο εγκληματίες και πολλά από αυτά τα οποία θα πω σε αυτό το σημείο έχουν καλυφθεί ιδιαίτερως από, το, από την πλευρά του Proof House. Τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται δεν είναι τα ημιαυτόματα όπλα, αλλά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στο υπάρχον σύστημα ε, νομοθεσίας και η ζήτηση για αυτά στους εγκληματικούς κύκλους χαρακτηρίζεται από την ανωνυμία τους και τη δυσκολία να εντοπιστούν και την ευκολία να μετατραπούν ε, και να αλλάξουν. Αυτά λοιπόν τα οποία είναι πιο εύκολο να μετατραπούν, αυτά θα έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Γιατί είναι έξω από το σύστημα. Ένα θέμα το οποίο μιλείς αναφέραμε ήδη είναι ότι κάτι το οποίο κάποτε ήταν ένα όπλο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο. Ισχύει εδώ. Ε, θα ήθελα να σας πω κάτι για την απενεργοποίηση όμως. Το πρώτο είναι τα όποια ε, κοινά χαρακτηριστικά και πρότυπα τα οποία θα ε, υιοθετηθούν ε, δεν θα πρέπει να έρχονται εις βάρος των εθνικών προτύπων, δεν θα πρέπει να είναι μια δικαιολογία για τα ε, πρότυπα υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό συμβαίνει, όπου οι άνθρωποι δεν βλέπουν την ανάγκη να τα απενεργοποιήσουν, τα απενεργοποιημένα όπλα ε, δεν είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τους ε, συλλέκτες, διότι προτιμούν να διατηρήσουν τα αρχικά χαρακτηριστικά των όπλων τους. Και δεύτερον, τα απενεργοποιημένα ε, τα στοιχεία των απενεργοποιημένων όπλων θα πρέπει να διατηρούνται διότι έχουμε περιπτώσεις όπου απενεργοποιημένα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί το οποίο σημαίνει ότι τα πρότυπα απενεργοποίησης δεν είναι ιδανικά. Οπότε θα πρέπει να έχουμε αυτά τα δεδομένα για την ειχνηλωσιμότητά τους. Επίσης πολλά δεν έχουν καταγραφεί αρχής εξ αρχής ως πολιτικά όπλα Είχαμε ακούσει, ακούσαμε περιπτώσεις όπου, άνθρωποι, όπου χρησιμοποιήθηκαν όπλα τα οποία έριξαν ε, άσφαιρα ε, και στη συνέχεια μετατράπηκαν. Και νομίζω ότι το βασικότερο εδώ πέρα είναι το οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε ε, όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν θα πρέπει να θεωρείται απομίμηση και αντίγραφο. Οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί θα πρέπει να αντιμετωπίζεται λοιπόν σαν όπλο ή ο ειδικό ε, προτείνει ότι λίγο πολύ το οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί, ε, οπότε η μείωση κινδύνου είναι να καταλάβουμε τι πρότυπα θα πρέπει να υπάρχουν σχετικά με το τι μπορεί να μετατραπεί εύκολα και πάλι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη κοινή κατανόηση σχετικά με το τι είναι ε, μετατρέψιμο και τι όχι και αυτό να το μετατρέψουμε σε εφαρμόσιμα πρότυπα και ε, η συζήτηση να περιλαμβάνει και τα ε, ουσιώδη συστατικά στοιχεία του όπλου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κρεπίνκο από την Europol. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ προτίμασα μία παρουσίαση. Αν όμω δεν μπορούμε να τη δούμε στι οθόνε, τότε μπορώ να κάνω και μια σύντομη παρέμβαση εκτό παρουσίαση. Ξεκινήσω λοιπόν με μια πολύ σύντομη παρουσίαση τη Europol για να αποφευθούν τυχόν παρανοήσει σε μελλοντικέ συζητήσει. Στη Europa λοιπόν έχουμε ως ε, σκοπό να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα τη συνοριακή του διάσταση. Και έχουμε και μια συγκεκριμένη τώρα ε, ομάδα που ασχολείται μόνο με τα πυροβόλα όπλα, την παρασκευή τους και την θέση τους σε εμπορία. Σε αυτά τα δύο χρόνια Βλέπουμε ότι η εντολή μας ήταν εξαιρετικά στενή και περιορισμένη. Τώρα την διευρύνουμε. Έχουμε και μικρά όπλα, πρόδρομες ουσίες. Έχω φτιάξει ορισμένες διαφάνειες για να σας δώσω ε, επιγραμματικά κάποιες εικόνες, αν και δεν έχουμε πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν. Έχω κάποια τεχνικά προβλήματα, συγγνώμη. Εντάξει. Έχετε λοιπόν μια επισκόπηση των υπόπτων που έχουμε εδώ πέρα στι βάσει δεδομένων μας. Βλέπουμε ότι κανένα κράτο μέλος δεν ε, έχει απαλλαγή από τα φαινόμενα αυτά. Ξέπερνα, μάλλον αφήνω κατά μέρο αυτά τα τμήματα γιατί έχουν ήδη αναφερθεί. Εγώ επικεντρώθηκα στα απενεργοποιημένα ή εκ νέου ενεργοποιημένα όπλα και έχω αφήσει κατά μέρο ε, τα στρατιωτικά όπλα που προκύπτουν από εμπόλεμε ζώνε και άλλες ε, κρίσιμες ζώνες. Αυτό που μας ε, προκάλεσε έκπληξη είναι ότι όταν είδαμε τα πρώτα στοιχεία από συγκεκριμένε εταιρείε από κάθε κρατημέλη, βλέπουμε ότι πουλάμε απενεργοποιημένα όπλα σε κάποιου αγοραστέ στη Δυτική Ευρώπη και αυτά τα όπλα που έχουν ήδη επενεργοποιηθεί ως αρχή επιβολής του νόμου ε, τα ανοιχνεύουμε και φτάνουμε και πάλι μέχρι την ε, εταιρεία και βλέπουμε ότι ήταν ε, απόλυτα νόμιμες αυτές ε, οι εταιρείες, κανένα πρόβλημα, αλλά βλέπουμε πώς ανέβηκαν οι πωλήσει της εταιρείας αυτής και πόσο δύσκολο ήταν για εμάς να δούμε ακριβώς τι έγινε με την αγοραπολισία, τα έγγραφα, ήταν όλα λίγο ε, σε μια γκρίζα ζώνη. Βεβαίως δεν θέλω να θίξω κανέναν ε, και πραγματικά Πιστέψτε με, εγώ δεν ε, θέτω αναμφιβόλο την χρήση των όπλων ή την αγοραπολισία των όπλων εν γέννη. Απλώς σας λέω ποια ήταν η εμπειρία μου όταν είδαμε με αυτά τα όπλα που θεωρούσαμε ότι εύκολα θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν εκ νέου και να χρησιμοποιηθούν ε, στο οργανωμένο έγκλημα και στην τρομοκρατία. Εδώ έχετε τις ε, παρτίδες που απεστάλησαν σε όλη την Ευρώπη, τις οποίες καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε. Και μετά συγκεντρώσαμε τα κράτη-μέλη και μοιραστήκαμε αυτέ τι πληροφορίε μαζί του. Και του ετέθησαμε να τα εξετάσουν. Γιατί όλα τα κράτη-μέλη που απευθύνονται σε εμά είπαν. Ναι, υπήρξαν κατασχέσει επανεργοποιημένων όπλων και μάλιστα από οργανωμένους εγκληματίες και όλοι είχαμε εκπλαγεί για το πώ αυτό ήταν δυνατόν. Εδώ έχετε μία εταιρεία που ε, δραστηριοποιείται συνήθως και κυρίως ε, στα άσφαιρα και οι δικές τους ε, πωλήσει έχουν ανέβει πάρα πολύ. Κλείνοντας, και να σας δώσω και χρόνο για ερωτήσεις αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της νόμιμης χρήσης των όπλων, Βεβαίω, ε, Θα ήθελα όμως να ζητήσω να υπάρξει μια πιο δομημένη δυνατότητα των αρχών επιβολή του νόμου να κάνει τη δουλειά τη ε, και σε ό,τι φορά την ε, εφαρμογή των νόμων αλλά και σε ό,τι φορά τις έρευνες. Όταν έχουμε έρευνες σχετικά με μια ομάδα που χρησιμοποιεί όπλα που έχουν αγοραστεί κατά τέτοιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. θεωρητικά τώρα θα έπρεπε να ξεκινάει η συνεδρία των συντονιστών. Δεν ξέρω αν σας πειράζει να καθυστερήσουμε τα 15 λεπτά έως και μισή ώρα. Εντάξει, θα δούμε. Συνεχίζουμε τέλος πάντων. Ερωτήσεις. Θα κάνω εγώ το πρώτο ερώτημα, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Από το αίτημα ε, που αναφέρθηκε να υπάρχει πρότυπο κανόνας για την μετατρεψιμότητα. Κατανοώ ότι είναι ζήτημα, αλλά υπό την ισχύουσα οδηγία που δεν προτείνει να τροποποιηθεί σε αυτό το σημείο, είναι σαφές το άρθρο 1, ότι ένα αντικείμενο θεωρείται πυροβόλο όπλο εάν υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του σε όπλο. Εάν λοιπόν κάτι μπορεί να μετατραπεί σε πυροβόλο όπλο, τότε θεωρείται όπλο. Και εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Είναι σαφές ήδη από το άρθρο 1 Κατανοώ λοιπόν την ανάγκη ύπαρξης ε, πολύ αυστηρών προτύπων για την επενεργοποίηση και ούτω καθεξής, αλλά σε ό,τι αφορά ε, τη δική μου θεώρηση του νόμου, ε, αυτή η εταιρεία στη Σλοβακία έτσι και αλλιώς ήταν παράνομη σαφώς, γιατί πολλούσαν αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε όπλα και έτσι η δραστηριότητα αυτή ήταν παράνομη αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα, αλλά θα δώσω το λόγο στην Άννα Μαρία. Ευχαριστώ πολύ, εν συντομία. Και εγώ πραγματικά έχω σοκαριστεί και λυπάμαι πάρα πολύ για τον τραυματισμό των τριών Βέλγων αστυνομικών. Έχουμε καλή ανάρρωση στους συναδέλφους σας. Θα ήθελα ε, να πω κάτι ε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ομοιότητας συμφωνώ, πρέπει να υπάρξει, να ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα στην οδηγία, ότι δεν είναι θέμα όψης και εικόνα, είναι θέμα ουσία. Ε, το βασικό μου ερώτημα όμω το απευθύνω στη Europol, γιατί αυτό που μα παρουσιάσατε μας προβληματίζει, γιατί δείχνει ότι είναι μια αυξητική τάση. Τι κάνετε λοιπόν εσείς γι' αυτό, θεωρείτε ότι η συνεργασία μεταξύ των μελών είναι επαρκής και ότι τα όσα υπάρχουν στην οδηγία αρκούν σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή πτυχή και, τα, και το φαινόμενο αυτό, τα νόμιμα όπλα να γίνονται παράνομα, το, το οποίο είναι και αυτό που μας απασχολεί. Πρώτα τα πλήρη μέλη της Επιτροπής, μετά τα πληρωματικά και μετά οι υπόλοιποι. Ανδρέας Σφόμπ. Παρακαλώ. Ich habe zwei Fragen. Zum einmal an den ähm, Ερωτήματα προς τον εκπρόσωπο της Βελγικής Αστυνομίας ο οποίος ε, ε, ήταν ιδιαίτερα κριτικός σχετικά με τα ε, πολεμικά όπλα, το οποίο στο γερμανικό δίκαιο συζητούμε ιδιαίτερο, και για το ότι κάτι δεν λειτουργεί ή όχι. Κάθε, όσον αφορά την οργάνωση ΦΑΤΣΕ, κάθε τόσο μιλάμε για αυτόματα και μη αυτόματα όπλα, θα μπορούσατε να πείτε για ποιο λόγο οι κυνηγοί χρειάζονται τέτοια όπλα. Καλδερά. Ευχαριστώ. Εντάχει. Ε, επειδή έχουμε εδώ αστυνομικούς από Βέλγιο, Γαλλία και από την Ιντερπολ, θέλω να θέσω μια σημαντική για μας ερώτηση. Κατά την άποψή τους, η ύπαρξη διαφορετικών νομοθεσιών στην Ευρώπη που μπορεί να επιβαρύνει τις δυνατότητες παρέμβασης διότι το ερώτημα που εμείς θέτουμε και δεν είναι θέμα της επικουρικότητας, αυτό είναι θέμα επιλογής των κρατών, το, είπο, το είπανε. Ε, οι ευρωβουλευτές πρέπει να ορίσουν κανόνες που σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να διευκρινίσουν την, ε, να διευκολύνουν τη δουλειά μας, γιατί είναι προφανές ότι καταλαβαίνω το δικαίωμα των ιδιωτικών ε, συμφερόντων, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το καθεστώς έτσι όπως έχει. Η αύξηση της ανάγκης ε, να συνεργάζονται οι αστυνομικές υπηρεσίες. Θα ήθελα λοιπόν να δώσουμε έμφαση στα διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια. Δημιουργούν πρόβλημα στην αστυνομία ή όχι. Um, you Uh, Ευχαριστώ. Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες οδηγίες, ε, μια από τα πιο αφιλεγόμενα στοιχεία είναι η απαγόρευση των ημιαυτομάτων που μοιάζουν με αυτόματα. Η ίδια η Επιτροπή λέει ότι η πρόταση δεν είναι ικανοποιητική και η πρόταση κατάργηση κάποιων εξωτερικών στοιχείων του όπλου θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση. Τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται σε εξάσκηση, σε πρακτική και σε σκοποβολή. Αυτό που κάποιοι τα θεωρούν στρατιωτικά στοιχεία είναι στοιχεία που βελτιώνουν την ακρίβεια και την εργονομία των όπλων που είναι σημαντικά για τους ε, αθλητικούς, ε, για, τους, ε, για το άτομο που χρησιμοποιούν τα όπλα για αθλητικές δραστηριότητες, όχι για τρομοκράτες η δυνατότητα να ε, περιοριστεί η δυνατότητα να περι, περιορισμός της δυνατότητας αυτός δεν ε, δίνει, ε, δεν δίνει αποτελέσματα. Αν δώσουμε κάποια ένδειξη ότι θα υπάρξει απαγόρευση του συγκεκριμένου όπλου μπορεί να αρχίσουν να αγοράζουν περισσότερα. Αυτό κάνει, συμβαίνει όταν αρχίζεις να, αγορα... να απαγορεύεις κάτι που είναι ελεύθερο. Ποια είναι η άποψή σας για τις προτάσεις ένα περίστροφο κατά την άποψή είναι περισσότερο επικίνδυνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο συχνά σε έγκλημα αν περιλαμβάνει ας πούμε στρατιωτικά χαρακτηριστικά όπως ε, ε, ε, σκανδάλι περιστρόφου στα σκανδάλι πιστολιού και επιπλέον τι είναι το ουσιώδες στοιχείο εδώ ο Γέντς Μπένσον Ευχαριστώ εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έχει εξαιρετικά αυστηρή νομοθεσία στον τομέα αυτό και δεν υπάρχει μεγάλη προσθέμενη αξία στην πρόταση επιτροπή. Κάτι σημαντικό είναι ωστόσο τα απενεργοποιημένα. Μπορεί να μου πούν αν το AK-47, το καλάστικο δηλαδή, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την απενεργοποίηση ή οποιοδήποτε στο πάνελ. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι κυνηγοί ή χρήστες όπλων για αθλητικούς σκοπούς θα επηρεαστούν από την, από την απαγόρευση αυτών των ημι, των ημι ε, αυτόματων που μοιάζουν με αυτόματο. Παρόμοια ερώτηση με αυτή που τέθηκε ήδη Ο εκπρόσωπος ε, από τη Λίμπη, ο κύριος Βαλέρα, η κυρία Βαλέρα, θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Αγγλικά θα μιλήσω, γι' αυτό βάλτε κανένα ακουστικό. Και λυπάμαι που δεν μπορούσα να είμαι εδώ συνολικά. Είχαμε μια σημαντική ψηφοφορία για την Τουρκία. Πήρε μια ώρα για να ψηφίσουμε. Το, εδώ το θέμα είναι δύσκολο και τεχνικά και ουσιαστικά. Τι σημαίνει ότι η Επιτροπή θέλει να απαγορεύσει, ας πούμε, θέλει να απαγορεύσει όλα αυτά τα όπλα η Επιτροπή. Ο συνάδελφος από την Φιλανδία μίλησε για τους γεμιστήρες ε, ένα θέμα που είναι πρόβλημα, ιδίω οι γεμιστήρε μεγάλη χωρητικότητα που χρησιμοποιούνται από λάθος χρήστε σε λάθος όπλα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Πώς μπορούμε να ε, διαχειριστούμε το θέμα των γεμιστήρων. Είναι θέμα επινσήμανσης μόνο. είναι η επισήμανση των γεμιστήων ως τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα ασφάλειας. Ευχαριστώ και θα θέσω άλλο ένα τελευταίο ερώτημα σχετικά με τους γεμιστήρες ε, και θα ήθελα να επαναλάβω και πάλι το σεβασμό μου ε, για την ε, βελγική αστυνομία και τις προσπάθειες ε, και το έργο που κάνουν ώστε να μας κρατήσουν όλους ασφαλείς. Όσον αφορά τους γεμιστήρες, κανένας δεν έθεσε το ερώτημα σχετικά με τις εκτυπώσεις 3D και την ικανότητα να, να δημιουργήσουμε πλαστό εξοπλισμό. Ίσως ε, θα ήταν λοιπόν εύκολο ε, να κάνουμε μια απομίμηση σχετικά με τους ε, γεμιστήρες. Θα πρέπει λοιπόν ε, ο έλεγχος κατ' εμέ δεν είναι λοιπόν ε, η καλύτερη προσέγγιση και δεν θα είναι πολύ εύκολο διότι είναι εύκολο να, το, να δημιουργηθεί απομίμηση. Δεν ξέρω λοιπόν ότι αν έτσι θα επιληθεί όντω το πρόβλημα. Ίσως η κυνηγητική οργάνωση μπορεί να βρει μια λύση να, υπάρχει, να υπάρχουν γεμιστήρες ε, που να έχουν μια περιορισμένη χωρητικότητα, όμως να τα αντιμετωπίζουμε ως ε, ουσιώδη συστατικά στοιχεία, κατά δεν φαίνεται ότι είναι η ιδανική λύση με βάση τα όσα άκουσα. Με ό,τι σειρά θέλετε, ίσως και αντίστροφα. Πρώτη η Europol. Καλή ιδέα, ευχαριστώ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε αρχικά ότι ε, τα απενεργοποιημένα όπλα ε, ε, σε περίπτωση που μπορούν να επανεργοποιηθούν τότε δεν θα πρέπει να θεωρούνται τέτοια. Επέλεξα το σλοβακικό παράδειγμα επίτηδες διότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους ε, σλοβάκους ε, συναδέλφους και η ανταπόκριση τους ήταν πάρα πολύ άμεση και προοδευτική ε, μπορώ να πω. Δεν είναι η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά οι εταιρείε τους εκεί αποτελούν τους μεγαλύτερους προμηθευτές στην Ευρώπη και έχουμε μια πολύ καλά οργανωμένη πανευρωπαϊκή ομάδα εργασίας που δουλεύει αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Τα καλά λοιπόν είναι και αυτά στη συγκεκριμένη κατηγορία λοιπόν. Ένα λεπτό για κάθε έναν από τους υπόλοιπους ομιλητές για να μιλήσει και η Κομισιόν. Θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν, λέει ο ομιλητής, συγκεκριμένα για τα πρότυπα της απενεργοποίησης ακόμα και αν το γράμμα του νόμου είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι η μετατρεψιμότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα τις βολές που γίνονται ε, σήμερα ε, χρησιμοποιούν μετατρέψιμα όπλα και παρόλο που η μετατροπή είναι ποινικό αδίκημα παρόλα αυτά θα πρέπει να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά του ε, στοιχείου που το κάνουν μετατρέψιμο είτε είναι τα υλικά από τα οποία αποτελείται το στοιχείο ή σχεδιαστικά πράγματα όπως είναι για παράδειγμα η κάνη θα πρέπει να εξετάσουμε αν ε, τα πρότυπα παραγωγής ε, μπορούν να επιτρέψουν ε, να χρησιμοποιείται νόμιμα το όπλο περιορίζοντας τη δυνατότητα μεταταψιμότητας διότι αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία οι αρχές αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αν ένα όπλο που ρίχνει άσφαιρα μπορεί να μετατραπεί τότε δεν θα πρέπει να το κατέχει κάποιος χωρίς να καταγράφεται. Αυτό όμω συμβαίνει καθημερινά. Άρα τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω αρχικά στο ερώτημα για ποιο λόγο οι κυνηγοί χρειάζονται μια αυτόματα όπλα. Διότι μπορούν να πάρουν πάνω από δύο σφαίρες και με βάση την οδηγία για το κυνήγι ε, πουλιών για παράδειγμα πτηνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, δύο, τρεις, ως και πέντε σφαίρες. Ή μπορεί να φτάσουμε και τις 20, τις 30 για το κυνήγι. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τέτοια, ε, τέτοιες σφαίρες μερικές φορές για επικίνδυνο ζώο, όπως είναι για παράδειγμα το κυνήγι αρκούδων στη Φινλανδία κάποια ζώα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα σε πυκνά δάση, χρειάζονται αυτά τα όπλα ε, και για, φυσικά για ηθικούς λόγους. Δεν θέλουμε να τραυματίσουμε το ζώο και να το αφήσουμε να υποφέρει, θέλουμε να το αποτελειώσουμε. Και τα όπλα, τα ημιαυτόματα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις γυναίκες, διότι είναι ένα εύκολο όπλο, μπορεί να το, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εύκολα τόσο οι γυναίκες αλλά ε, και ε, κυνηγοί που έχουν κάποια αναπηρία. Τώρα πόσοι κυνηγοί ε, αλλά και αθλητές θα επηρεαστούν δεν έχω έναν ξεκάθαρο αριθμό. Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί φοβάμαι από την Κομισιόν. Και τέλος το ερώτημα σχετικά με τους γεμιστήρες. Πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση η κυρία Φόρτ τόνισε ότι δεν αποτελεί ε, ουσιώδες θετικό του όπλου και γι' αυτό το λόγο θα προτείναμε να μην υπάρχει ε, χαρακτηρισμός. Όμως αν υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί για την ε, κατοχή, τότε θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε την εναλλακτική του να έχουμε μονάχα, ε, να, να, να, έχει τη δυνατότητα να το αγοράζει αυτό μονάχα κάποιος που έχει αρκετές ε, πιστοποιήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Στάσεν, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εντάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κάποια ουσιώδη στοιχεία. Βεβαίως και η προτεραιότητα για όλους είναι η ασφάλεια. Πολλοί ομιλητέ επέμειναν στη σημασία της συχναλησιμότητας, της ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά βεβαίως είναι εξαιρετικά ουσιώδη, όμως όλα αυτά θα λειτουργήσουν μόνο αν έχουμε δεδομένα στη διάθεσή μας. Μόνο δηλαδή εάν οι κάτοχοι των όπλων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία τα μουσεία, οι συλλέκτες που σήμερα δεν υπάγονται στην οδηγία. Εάν παραμείνουν εκτός, τότε το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών ε, δεν έχει νόημα, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Η χνελεθμότητα είναι σημαντικό σημείο και στο πλαίσιο της εγκληματικής δραστηριότητα, γιατί έτσι ανεβαίνουμε στην αλυσίδα και βλέπουμε από πού προήλθε η βασική προτεραιότητα δεν είναι να βρούμε ποιος διέπραξε το έγκλημα, είναι να αποτρέψουμε το έγκλημα. Για τα μουσεία, πολύ σύντομα. Κάποια μουσεία είναι πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως εδώ στο πάρκο στην Καντνέχ. Αυτά τα μουσεία έτσι κι αλλιώ δεν ε, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή οδηγία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για τι αντίκε και αυτά τα όπλα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή οδηγία βάσει και ε, τη ε, συνθήκη του, του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν για τα μουσεία. Μένει λοιπόν μόνο το ζήτημα των ε, σύγχρονων όπλων. Εδώ συμφωνούμε όντως ότι τα μουσεία που είναι ανοιχτά προς το κοινό θα, όντως ε, εκπληρώνουν και έναν κοινωνικό ρόλο. Πρέπει να υπάρχει, υπάρχει λοιπόν ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, όμως ε, είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές συλλογές. Δεν βλέπουμε γιατί θα πρέπει ο συλλέκτης να έχει το δικαίωμα να έχει στο σπίτι του στρατιωτικά όπλα και μάλιστα ενεργά θεωρούμε ότι οι συλλέκτες θα πρέπει να ε, υπάγονται στις ίδιες ε, προϋποθέσεις με ε, τον αθλητικό, την αθλητική σκοποβολή και ερευνητική σκοποβολή. Σε ό,τι αφορά τους κυνηγούς, συνήθως έχουν δικαίωμα για 4-5 σφαίρες. Επομένω, δεν τίθεται το ζήτημα της ίδιας προβληματικής του ημιαυτομάτου. Είναι βάση λοιπόν της λειτουργίας. Λοιπόν, για την ε, σκοποβολή είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Όντως ε, το Β7 η κατηγορία αυτή δεν είναι σαφής, πρέπει να δούμε τα κριτήρια. Για την κατηγορία Β7 λοιπόν υπάρχουν όμως και Καλάσνικοφ στην κατηγορία Β7, τα οποία είναι σαρδιτικά όπλα που έχουν ως στόχο να σκοτώσουν, όχι ε, τη σκοποβολή. Έχουμε τα R15 που είναι ε, το μικρό αδερφάκι του M16 και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να απογορευτούν στο πλαίσιο της οδηγίας. Τελευταίο στοιχείο και θα μείνω εδώ. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τα αυτόματα και μη αυτόματα, άκουσα πολλές προτάσεις που λένε ότι πρέπει να έχουμε κριτήρια ε, για τη μετατροπή σε αυτόματα. Για μένα δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση, γιατί όλες αυτές ε, ε, οι μαζικές δολοφονίες που είδαμε έγιναν με μη αυτόματα όπλα. Η ε, το ερώτημα που έθεσαν οι δύο συνάδελφοι εδώ μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατηγορία Β7 αυτή τη στιγμή που είναι νόμιμη και ε, υπόκειται σε αδειοδότηση. Επομένως θεωρούμε ότι γνωρίζουν οι αρχές πόσα τέτοια όπλα υπάρχουν λογικά. Ε, πόσα υπολογίζετε ότι είναι αυτά τα όπλα, πού θα απαγορευτούν και ποια είναι η απάντησή σας ως προς τα αιτήματα αποζημίωσης. Αυτό ήταν το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα όπλα της κατηγορίας Β7 έχουν λάβει άδεια και έτσι πόσα θα απαγορευτούν. Και τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις. Ο ακριβή αριθμό δεν είναι γνωστό. Έχουμε ρωτήσει κάποια τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, όχι από κακή βούληση των κρατών, αλλά από τον κακό ορισμό της οδηγίας για το πεδίο εφαρμογή. Άρα θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα τι εννοούμε με τον όρο όπλα προς απαγόρευση για να γίνει κατόπιν ο εντοπισμός. Αυτά δεν, δεν υπάρχουν στοιχεία αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, αποζημίωση συνδέεται με την πρώτη. Εφόσον δεν ξέρουμε πόσα όπλα υπάρχουν, το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπολογιστεί. Να υπολογιστεί επιπλέον. Πριν μιλήσουμε για αποζημίωση πρέπει να εξετάσουμε τυχόν μεταβατικά μέτρα που μπορεί να αποφασίσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που θα επιτρέψει την αποφυγή, την αποφυγή πιθανώς Προφανώ τη δυνατότητα ή τη υποχρεώση αποζημίωση. Okay. Δεν θέλω να κόψω κάποιον που θέλει να λάβει απάντηση, αλλά έχετε και το χρόνο. Νομίζω ότι απαντήθηκαν τα ερωτήματα που τέθηκαν. Είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν απαντήθηκε το ερώτημά σας κύριε Φέλνερ αυτό είναι ενδιαφέρον από μόνο του, αλλά άκουσα δύο, συναδε, δύο σχόλια. Αν υπήρχε σύνδεση μεταξύ αυτομάτων όπλων που χρησιμοποιήθηκαν παράνομα και αν είχαν στατιστικά γι' αυτό. Δύο συνάδελφοι το είπαν και θα ήθελα να ακούσω, να απαντάει η Επιτροπή τέλο πάντων. Τι θέλουν να διορθώσουν εν πωλής Κομισιόν. Το ρώτησαν συνάδελφοι. Δυστυχώς υπάρχει σύνδεση μεταξύ ήμι αυτομάτων και εγκλημάτων. Οι 77 νέοι που σκοτώθηκαν στην οδηγία σε μια κατασκήνωση με ημιαυτόματο που είχε όμως νόμιμα στη διάθεσή του υπήρξε μια σφαγή στο, σε ένα σχολείο στην Βρετανία, στη Γερμανία, στο Γενικό Συμβούλιο των Ντεσέν στο Παρίσι. Υπάρχουν πολλές δυστυχώς περιπτώσεις ε, ατόμων με ημιαυτόματα που πολλές φορές τα είχαν παράνομα στα χέρια τους. Νόμιμα στα χέρια τους. Να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες θα υποβάλουμε τοπολογίες για την έκθεση. Υπάρχουν κάποια εκκρεμή θέματα ακόμα που είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουμε εγγράφος και με ψηφοφορία. Ευχαριστώ.